Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ γιατί έχουμε καθυστερήσει πολύ και δεν θα ήθελα η δημοσία κρόαση της Ούρσουλας να μην λάβει την προσοχή που της αξίζει. Ήδη χάσαμε μισή ώρα από το χρόνο της δημόσια και πραγματικά ζητώ συγγνώμη από όσους περίμεναν έξω από την αίθουσα. Πάντως ο στόχος της ε, απογευματινής ακρόασης είναι να συνεχίσουμε τη συζήτηση ε, του θέματος πραγματεύεται στην γραμματότησή της Ιούρσουλα Λαγκάτσεκ Γκάτσεκ ε, με τα προβλήματα δηλαδή και τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Δώσουμε το λόγο στην εισηγήτρια της γνωμοδότησης, στον Επίτροπο Μπαρό και θα ακούσουμε πώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιμετωπίζει τους κανόνες που έχουν στόχο την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας καθώς και τις βελτιώσεις ε, που θα λάβουν χώρα στον τομέα αυτό που είναι δυνατόν να υλοποιηθούν. Επίσης ε, ε, θα έρθει σε λίγο και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής, ο κύριος Διαμαντούρος, που θα μας ενημερώσει για τις πιο συνηθισμένες αιτιάσεις και αναφορές των Ευρωπαίων πολιτών στην προσπάθειά του να ασκήσουν τα δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Θα ακούσουμε επίσης και εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων. Ο Πολωνός ε, υφυπουργό ε, Πιότρ Σταχάντσικ ε, δυστυχώς κολλείεται, αντικαθίσταται από τον κύριο Ματέου Σόρα. Δεν θα χρονοτριβήσω άλλο, θα δώσω αμέσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον Ζακ Μπαρό, για την εισαγωγή του και κατόπιν στη συντάκτη της γνωμοδότησής μας, την κυρία Ούρσουλα Γκάτσεκ. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ κύριε Γκάτσεκ και σας ευχαριστώ όλους θερμά για την παρουσία σε αυτή τη δημόσια ακρόαση. Η αυτή με θέμα την Ευρωπαϊκή Θεγένεια νομίζω ότι πέφτει την κατάλληλη στιγμή γιατί εκπονούμε το πρόγραμμα της Στοκχόλμης και θέλουμε να δώσουμε αυτό, σε αυτό το το, την, αυτή την έννοια τη ευρωπαϊκή ηθαγένεια σε ένα πιο συγκεκριμένο περιεχόμενο, να το δώσουμε σάρκα και οστά. Τι νόημα να δώσουμε σήμερα την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Από νομική άποψη, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι κυρίως ένα καθεστώ. Πρώτα απ' όλα, ένα καθεστώ. Ένα καθεστώ που επιτρέπει στου υπηκόου των κρατών μέλων να λάβουν άσχετα από την υπηκότητά τους την ίδια ε, νομική μεταχείριση όπου και αν βρίσκονται. Οπότε το καθεστώ αυτό απαρτίζεται από συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσει που προσδιορίζονται στη συνθήκη. Ελευθερία διακίνηση εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε στις ε, δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές σε ένα άλλο κράτος μέλος. Δικαίωμα προξενικής προστασίας δικαίωμα αναφοράς και υποβολή αιτίας προς τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, δικαίωμα να αποταθεί ο πολίτης στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή γίνει όμως είναι και μία έννοια με μεταβλητό περιεχόμενο μερικές φορές. Χάρη σε αυτή την έννοια θα έχουμε μία χρήσιμη συζήτηση για τη σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους πολίτες της. Βέβαια, η έννοια του Ευρωπαίου πολίτη είναι μάλλον ε, ένα φανταστικό ε, μόρφωμα. Χρησιμοποιείται πολλές φορές με αφηρημένο τρόπο και για διάφορους, πολλούς και διάφορους σκοπούς. Τι θα πρέπει λοιπόν να γίνει για να δώσουμε μια νέα όθηση στην πολιτική Ευρωπαϊκή Συνταγένεια της Ένωσης. Θα με ρωτήσετε όλοι θα πρέπει καταρχήν να ξεκινήσουμε ευρύτατες διαβουλεύσεις προκειμένου να συγκεντρώσουμε πληροφορίες για τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Έτσι θα μπορούσαμε να υποβάλουμε νέες προτάσεις με βάση τη συλλογή όλων αυτών των στοιχείων. Γιατί πρόκειται να συντάξουμε και νέα έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Επίσης θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε την ε, έμπρακτη άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θα πρόσθετα και τρεις άλλους άξονες. Η γνώμη του Ευρωπαίου πολίτη είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλίσουμε τη σωστή εφαρμογή των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια ελεύθερη διακίνηση, όπως σας είπα και προηγουμένως, δικαίωμα εκλέγει και εκλέγεστε. Θα πρέπει να διαφερθούμε ε, για τα διάφορα στάδια της ζωής του πολίτη, από την γέννησή του μέχρι το θάνατό του, περνώντας από το γάμο, τα παιδιά, την παιδεία, τη σύνταξη, τη μετακίνησή του στις διάφορες χώρες Ένωσης. Έχουμε το πρόγραμμα δράσης για την προξενική προστασία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό είναι το θέμα της, ε, του βίου του πολίτη. Μετά έχουμε το θέμα της συμμετοχής του πολίτη στον βίο της Ένωσης. Συμμετοχή στην ε, δημοκρατική συμμετοχη στην, Ευρωπαϊκή Ένωση, προώθηση του, του δικαιώματο συμμετοχή στι ε, δημοτικέ και ευρωπαϊκέ εκλογέ. Ένα κεκτημένο δικαίωμα που δεν χρησιμοποιείται. 12% των ε, ε, πολιτών έχουν εγγραφεί στι τελευταίε ευρωεκλογέ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Εργασίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την αναθεώρηση της πράξης του 1996 και αν γίνει αυτή η αναθεώρηση θα πρέπει να αναθεωρήσουμε και τη σχετική οδηγία που προσδιορίζει τους όρους εφαρμογής. Να ξεκινήσουμε μια μελέτη για την χαμηλή συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν σε χώρα που δεν είναι η δική τους για να αντιληφθούμε ποιο, πώς δικαιολογείται αυτό το χαμηλό ποσοστό συμμετοχής. Να γίνουν μελέτες συμβατότητας ε, των ε, εθνικών νομοθεσιών με την ε, πράξη του 1996 και από τα απορίσματα αυτής της μελέτης που θα περιμένουμε την άνοιξη του 2009 θα καταλήξουμε σε κάποιες συστάσεις. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε το δίκτυο πολίτες χωρίς σύνορα οι πολίτες που διαμένουν σε χώρα πλήν της δικής τους πατρίδας θα πρέπει να γίνουν κινητήρες μοχλός ε, του βίου της χώρας φιλοξενίας και να συμμετέχουν στις κοινωτικές πολιτικές. Μήπως λοιπόν θα πρέπει να ενθαρρύνουμε τη θέσπιση ενός δικτύου που θα φέρει σε επαφή ε, τα διάφορα μέλη της κοινωνίας των πολιτών ε, και στη χώρα, συμμετοχή, χώρα υποδοχής. Επίσης, συμμετοχή ε, και των παιδιών. Το Φόρουμ των Δικαιωμάτων των Παιδιών εκπονεί μια μέθοδο προκειμένου να συμμετέχουν και τα παιδιά στην εκπόνηση των πολιτικών της Ένωσης. Συμμετοχή στην πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για τον πολίτη. Έχουμε τα νέα δικαιώματα που προβλέπει η Δίκη τη Λισαβόνα και που επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο τουλάχιστον πολίτε τη Ένωση από διάφορε χώρε να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικέ προτάσει Βεβαίω, οι διαδικασίες και οι όροι εφαρμογή αυτού του νέου δικαιώματος ε, θα απαιτήσουν την ε, θέσπιση ενός κανονισμού. Τρίτο θέμα. Μην ξεχνάτε το προηγούμενο δύο ήταν τι νόημα θα δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και το δεύτερο, ποιε είναι οι συγκεκριμένε εφαρμογέ αυτή τη Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Το σημείο 3 είναι πώ θα συνδυάσουμε την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια με την εθνική υπηκότητα, γιατί κάποιο θα πρέπει να είναι υπήκο μια χώρας για να έχει και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Το θέμα τη διασύνδεση τη Ευρωπαϊκή ηθαγένεια με τη εθνική υπηκότητα δεν έχει συζητηθεί διεξοδικά. Βέβαια το θέμα τη υπηκότητα άπτεται της ε, αρμοδιότητα ε, των κρατών μελών και που θα πρέπει να ασκείται στα πλαίσια φυσικά του σεβασμού του κοινοτικού δικαίου. Οι διαφορές όμως ε, μεταξύ των εθνικών συστημάτων για τη χωρίση υπηκότητας έχουν ε, και κοινοτική επίπτωση. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ενημέρωση από τα κράτη-μέλη ε, όταν αποκτούν την υπηκότητα για τα δικαιώματα που δημιουργεί αυτή και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Μερικές φορές με ρωτούν οι πολίτες δεν θα ήταν σκόπιμο να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα, ένα ευρωπαϊκό δελτίο ταυτότητας. Βέβαια κάποια κράτη είχαν προβλήματα με την πρόταση αυτή, αλλά γιατί να μην εξετάσουμε και αυτό το ενδεχόμενο. Πάντως έχω εμπιστοσύνη στο καταπληκτικό σχέδιο έκθεση κυρίας Ουρσούλα Γκάτσεκ που θα σας ε, επιτρέψουν να εξετάσετε ποιες δράσεις θα πρέπει να εφαρμόσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δώσει νόημα αυτό περιεχόμενο σάρκα και οστά στην έννοια της Ευρωπαϊκής αγένειας. Ο Αγίος Παύλος είπε «Είμαι Ρωμαίος πολίτης». Και αυτό έχει νόημα. γιατί ως Ρωμαίος πολίτης δεν θα την πετοπιστεί ως οποιοδήποτε πολίτης. Εμείς δεν έχουμε φτάσει βέβαια εκεί, αλλά γιατί να μην φτιάξουμε την Ευρωπαϊκή Θαγένεια που δεν θα έρχεται σε αντίθεση ε, με την εθνική υπηκότητα, αλλά θα τη συμπληρώνει αυτή την εθνική ηθαγένεια και υπηκότητα. Έτσι θα επιτρέψουμε στα παιδιά και τους νέους της Ευρώπης να καταλάβουν την τύχη που έχουν να είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ε, merci, Σας ευχαριστούμε κύριε την Πρόεδρε. Ευχαριστώ Ζακ. Γνωρίζω ότι θα πρέπει να φύγετε σε λίγο γιατί σας περιμένει ο κύριος Μπρούγκερ για να δώσετε κοινή συνέντευξη τύπου. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέντευξη τύπου. Θα δώσω λοιπόν το λόγο αμέσως στην εισηγητριά μας, την Ούρσουλα Γκάτσεκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Καταρχήν ως εισηγήτρια πρέπει να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω τόσο εκπροσώπους των ε, πολιτών της Ευρώπης εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για ηθαγένεια, για τη σημασία που έχει η ηθαγένεια στους πολίτες της Ευρώπης χωρίς εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων εδώ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είστε εδώ λοιπόν. Όταν άρχισα να εργάζομαι πάνω στην έκθεση δεν υποπτευόμουν ότι θα προκαλούσε τόσο ενδιαφέροντα και αντιτιθέμενα σχόλια στην Πολωνία γιατί ήταν το αντικείμενο έντονων συζητήσεων σε πολλά φόρα του διαδικτύου. Παρακολούθησα τις ε, αντιπαραθέσεις με ενδιαφέρον γιατί με έκπληξη διαπίστωσα ότι ήταν πολύ λίγα γνωστά σχετικά με τα δικαιώματα του Ευρωπαίου πολίτη αλλά και ότι δημιουργούσε έναν παράξενο φόβο ότι η εθνική ηθαγένεια δηλαδή θα αντικατασταθεί από μια μυθική ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Τους τελευταίους μήνες λοιπόν τους πέρασα στην πατρίδα μου εξηγώντας ότι αυτό είναι κάτι πρόσθετο και θετικό και όχι εναλλακτικό. Δεν υπάρχει μυθική ευρωπαϊκή ηθαγένεια που δεν εδράζεται ε, στέρεα στην εθνική νομοθεσία αλλά η συζήτηση που παρακολούθησα στα βήματα του ίντερνετ μου έδειξαν και που εξέφρασαν άποψη οι πολίτες εκεί ότι αυτά όλα δεν ήταν ξεκάθαρα σε πολύ κόσμο. Χαίρομαι πολύ που είχα τη δυνατότητα να εργαστώ πάνω στην έκθεση αυτή. Όπως γνωρίζετε, καλύπτει μία περίοδο κατά την οποία άλλαξε δραματικά η Ευρώπη, δηλαδή από την 1η Πρώτου του 2004, όπου η Ευρωπαϊκή ε, πρώτη του 2004, με συγχωρείτε, ε, όταν προσχώρησαν νέα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα τα κράτη της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης. Οι πολίτες της παλιάς Ένωσης ε, άρχισαν να ε, ε, ασκούν τα δικαιώματα αυτά ε, δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης κλπ. Όλα αυτά όμως δημιουργήσαν και πρακτικά καθημερινά προβλήματα στους πολίτες καθώς ε, μετακινούνταν από τη μία χώρα στην άλλη με τις διαφορετικές νομοθεσίες ε, δικαιικά συστήματα, προβλήματα νομολογίας, είχαν πολλά προβλήματα καθημερινά με δικαιώματα συνταξιοδότησης, ε, υπηρεσίες ε, υγείας, ε, διαζύγια, γάμοι. Είχαμε πολλά προβλήματα σε όλους αυτούς τους τομείς λόγω της επιθυμίας άσκησης των δικαιωμάτων που υφίσταντο. Πολλά από τα θέματα λοιπόν που μας απασχολούν στην έκθεση και στη συζήτηση ελπίζω επικεντρώνονται σε αυτά τα πρακτικά ζητήματα. Χαίρομαι πολύ που ο Επίτροπος ανέφερε κάτι που εγώ θεωρώ από ε, τα πιο σημαντικά στοιχεία της ε, συνθήκης της Λισαβόνας, η πρωτοβουλία του ενός εκατομμυρίου υπογραφών. Πολίτες που θεωρούν ότι η φωνή τους ε, γίνεται ακουστή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αν όμως η Ευρωπαϊκή, η Ένωση της Λισαβόνας ε, θα παγώσει μακροπρόθεσμα, τότε ε, δεν θα αξιοποιηθεί αυτή η πρωτοβουλία. Όποια για είναι η τύχη της συνθήκης της Λισαβόνας και πραγματικά προσεύχομαι να επιτύχει και να κυρωθεί, αλλά ε, τουλάχιστον αυτή η πρωτοβουλία δεν θα έχει χαθεί. Ε, θα μιλήσουμε για την προξενική προστασία και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών να προστατεύονται από το διπλωματικό και προξενικό προσωπικό των κρατών μελών, αν βρεθούμε σε κάποια δυσκολία ε, σε περιοχή όπου δεν υπάρχει εκπροσώπηση της χώρας μας. Αυτό το εγγυάται, το διασφαλίζει η συνθήκη. Είδαμε όμως ακόμα και από τις εμπειρίες των μελών της Επιτροπής αυτής ότι όταν περάσουμε στα πρακτικά ζητήματα της καθημερινής πραγματικότητας ε, διαφοροποιούνται τα πράγματα. Ένας συνάδελφος πρόσφατα ε, ήταν επικεφαλής της ε, αντιπροσωπείας του Μομπάι. Ξέρετε το μεγάλο ε, ατύχημα εκεί. Πολλοί στη, στη Μομπάι. Πολλοί ε, ευρωβουλευτές όπως και πολίτες Ινδοί βρέθηκαν να απειλούνται σε ό,τι φορά τη ζωή τους με τις πιτζάμες στο ξενοδοχείο και έπρεπε να βοηθηθούν από οποιοδήποτε προξενείο ήταν εκεί αν ε, ε, οι ευρωβουλευτές είχαν τέτοιο πρόβλημα στις δικαιωμάτων, ε, πόσο μάλλον ένας απλός πολίτης. Και αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν που το εξετάζομαι πολύ προσεκτικά. Επίσης με χαρά ε, βλέπω στην έκθεση αυτή ότι ήδη παρακολουθούμε εκ του σύνεγγις και επανεξετάζουμε και αναθεωρούμε τα διάφορα προγράμματα που ήδη υπάρχουν, έχουν θεσμοθετηθεί για να βοηθηθούν οι πολίτες να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Πολίτες ε, που για παράδειγμα βρίσκονται μεταξύ δύο δικαιικών συστημάτων και μετά έχουν και το γλωσσικό εμπόδιο να αντιμετωπίσουν. Πολύ συχνά λοιπόν δεν ξέρουν πού να απευθυνθούν είναι μακριά από τη χώρα τους, βρίσκονται σε μια άλλη χώρα, υπάρχουν προβλήματα ε, ε, μετάβασης από τον ένα οργανισμό στον άλλον, προβλήματα τοπικής αυτοδιοίκησης ακόμα έχουν πολύ δρόμο να κάνουν μέχρι την επίλυσή τους. Χαιρόμαστε που υπάρχουν προγράμματα, αλλά θα πρέπει να δοθεί ε, έμφαση στα προγράμματα αυτά έξω από το κλίμα των Βρυξελών για να μετατεθεί η έμφαση εκεί που αντιμετωπίζονται τα προβλήματα. Θα πρέπει με την έκθεση αυτή η αντίληψη περί ε, ιδιότητα του πολίτη να γίνει ορατή και κατανοητή από τους ίδιους τους πολίτες. Θα πρέπει λοιπόν εμείς ως θεσμικά όργανα, ως βουλευτές, ως μέλη της Επιτροπής, του Συμβουλίου, θα πρέπει να δούμε οι επικείμενες ε, ευρωεκλογές του Ιουνίου, όπως ο Επίτροπος είπε πολύ ε, σωστά, αυτές οι εκλογές χαρακτηρίζονταν από χαμηλή συμμετοχή στις εκλογές όχι από τους ανθρώπους που ψηφίζουν σε μια ξένη χώρα που δεν είναι υπήκοοι, αλλά είναι συμμετοχή χαμηλή ακόμα και στους επικόους μιας χώρας. Ίσως λοιπόν ε, αυτή η χαμηλή ε, συμμετοχή ε, να πρέπει να μας αφυπνήσει με δεδομένα τα αποτελέσματα των δημοψήφισμάτων, Ιρλανδία κτλ. Περνάνε τα μηνύματά μας, είναι σημαντικά τα μηνύματα που απευθύνομαι και ασχολούνται με τα θέματα που απασχολούν καθημερινά τους πολίτες. Ε, χαίρομαι πολύ που βλέπω εδώ εκπροσώπους κυβερνήσεων, μη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή, αλλά κυρίως με ενδιαφέρει να ακούσω τη δική σας τη φωνή γιατί ακόμα είναι ε, υπό επεξεργασία η έκθεση. Η προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών στην έκθεση αυτή λίγη αύριο. Αν λοιπόν μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, βρείτε κάποιον φιλικό ευρωβουλευτή που ε, θα τίνει ευήκον ους, μέχρι αύριο το μεσημέρι έχετε τη δυνατότητα να έρθετε σε επαφή και να συμβάλλετε στη διαμορφωσή των τροπολογιών. Euh, Σας ευχαριστώ ήταν πολύ συγκροτημένη και τεκμηριωμένη παρουσίαση αυτή της έκθεσής σου. Σε ευχαριστούμε θερμά. Θα ακούσουμε τώρα μία ανακοίνωση του κυρίου Ματέου Σόρα, που είναι διευθυντής του Τμήματος Ιθαγένειας και Παναπατρισμού στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας. Θα μας μιλήσει λοιπόν ο κύριος Σόρα για το τι προβλήματα Ιθαγένειας ανακύπτουν στην Πολωνία, ιδιαίτερα ε, υπό το πρίσμα μιας χώρας που πρόσφατα εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ακούσουμε λοιπόν τώρα τον εκπρόσωπο της ε, πολωνικής κυβέρνησης, τον κύριο Ματέους Σόρα. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε πρόεδρε, αξιότιμη κυρία εισηγήτρια, κυρίες και κύριοι. Το θέμα της ε, σημερινής δημόσιας ακρόασης είναι η πραγματοποίηση μιας αντικειμενικής αξιόλογης της πέμπτης ανακοίνωση Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά την 1η Πρώτου 2004 ε, μέχρι το 2007 και το άγραφο εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνει πληροφορίες σε σχέση με τα παραρτήματα 1, 2, 3 και 7 της έκθεσης αυτής. Η αξιολόγηση γίνεται και στα πλαίσια μια πρόταση ε, ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με θέμα το πρόβλημα και, τα προβλήματα και τι προοπτικέ ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, η έκθεση αυτή θα εκπονηθεί από την κυρία, από την Ούρσουλα Γκάτσεκ και μιλάει για τις ελευθερίες ε, και τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών στον Ευρωπαϊκό Χώρο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας. Όλα αυτά τα έγγραφα είναι πολύ σημαντικά και δείχνει την μέρημνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη και ενίσχυση της σημασίας των θεσμικών οργάνων στα μάτια του Ευρωπαίου πολίτη. Αυτά τα θεσμικά όργανα θα πρέπει να διαδραματίσουν ε, σημαντικό ρόλο στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ε, ολοκλήρωσης. Το θέμα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας συνδυάζει την ε, ε, συνέχιση της παραδοσιακής έννοιας της ηθαγένειας ως δεσμού νομικού που συνδέει τον άνθρωπο με το έθνος και σε συνδυασμό με την ευρωπαϊκή διάσταση. Όπως φαίνεται στα κοινοτικά ε, έγγραφα, για πρώτη φορά η δήλωση για την ευρωπαϊκή ταυτότητα που δέχτηκαν η αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων το 2003 στην Κοπεχάγη είναι πολύ σημαντική. Βέβαια, ο διαχωρισμός ε, μάλλον η Χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δείχνει πόσο σημαντικό είναι να αναγνωρίσουμε το δικαίωμα της ηθαγένειας ως θεμελιώδης δικαίωμα ανθρώπινο. Αυτό φαίνεται σε διάφορα ε, διεθνή έγγραφα και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση ε, του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, του 1979. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό αυτό το θέμα της ηθαγένειας και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας. Γιατί έχουμε έναν θεσμό εσωτερικού δικαίου και ένα θέμα παραδοσιακού κοινοτικού δικαίου, αλλά και θέμα διεθνούς δικαίου και κοινοτικού δικαίου. Θα πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη ότι με βάση το άρθρο 8 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφέρθηκε πολίτης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πάντως ε, περίεργο ότι δεν έχουμε στο ίδιο, στην ίδια αυτή συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτήν την αναφορά, αλλά στην ίδια τη συνθήκη της ε, ε ίδρυσης της Ένωσης. Η συνθήκη του Άμστερνταμ επίσης αναφέρει ότι ε, η ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν αντικαθιστά, αλλά συμπληρώνει την εθνική ηθαγένεια. Από τους ορισμού αυτούς μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η έννοια τη Ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν έχει καμία πρόθεση αντικατάστασης της εθνικής ηθαγένεια στα κράτη-μέλη. Είναι δυνατή λοιπόν η συνύπαρξη και των δύο ηθαγενειών, τη Ευρωπαϊκή και τη Εθνική από την άποψη των δικαιωμάτων του πολίτη θα πρέπει, όπως εγγυάται στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, αλλά και στη συνθήκη του Μάστριχτ και στη συνθήκη του Άμστερνταμ, η έννοια της ευρωπαϊκής ηθαγένειας δεν στηρίζεται σε, μια λίγο, σε ένα λίγο πολύ επίσημο ορισμό, στηρίζεται περισσότερο σε ένα κατάλογο δικαιωμάτων που ε, μπορεί να τα ασκήσει κάποιος που φέρει την, ανθρώπινη, την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Επίσης, ε, τέτοιου είδου δικαιώματα κατοχυρώνονται και προηγουμένως στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο, πριν ακόμη προταθεί έννοια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Για παράδειγμα, έχουμε δικαιώματα όπως το δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης ε, και εγκατάστασης ε, στην επικράτεια μιας χώρας μέλους ή το δικαίωμα υποβολής αναφοράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κυρίε και κύριοι, ο κατάλογο των δικαιωμάτων που συνδέονται με την ευρωπαϊκή Ιθαγένεια δεν είναι ένα εξαντλητικό κατάλογο δικαιωμάτων. Γιατί η συνθήκη του Άμστερνταμ αναγνωρίζει το δικαίωμα κάθε πολίτη τη Ένωση να αποτανθεί στα βασικά θεσμικά όργανα τη Ένωση και μάλιστα στη μητρική του γλώσσα. Επίση, δημιουργείται υποχρέωση του θεσμικού οργάνου να απαντήσει στην ίδια γλώσσα έχουμε κατοχυρώσει το δικαίωμα πρόσβασης ε, του πολίτη στα έγγραφα του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής. Μην ξεχνάτε και την ε, νομοθετική διακήρυξη του άρθρου 22 της Συνθήκης Ίδρυσης Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αναφέρεται ότι το Συμβούλιο μονομερώσει μετά από αίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συμπληρώσει ή να βελτιώσει τα δικαιώματα ε, των κρατών μελών, των πολιτών, όπως προβλέπονται από την Εθνική Νομοθεσία. Βέβαια τα, τα θεσμικά όργανα φαίνεται ότι δεν έχουν εξαντλήσει ακόμα αυτά τα δικαιώματα που κατοχυρώνονται από την ίδια τη συνθήκη. Μην ξεχνάτε ότι σε όλα τα έγγραφα που προανέφερα ε, θα μπορούσαμε ήδη να προτείνουμε κάποιες διατάξεις που να ενισχύουμε ή να συμπληρώνουμε τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Για παράδειγμα, στο σημείο 1 του σχεδίου ψηφίσματος της κυρίας Ούρσουλας Γκάτσεκ αναφέρεται η προετοιμασία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαφανής, διαφανούς διαδικασίας για την πρωτοβουλία αυτή των πολιτών και κατανοητής διαδικασίας. Σίγουρα αυτή η σύσταση είναι πολύ σημαντική. Από πρακτική άποψη βέβαια, η ελεύθερη διακίνηση και εγκατάσταση προϋποθέτει μία ενίσχυση. Γι' αυτό και στο σημείο 8 η κυρία Ούρσουλα Γκάτζεκ προτείνει η έννοια της ηθαγένειας να περιλάβει την αρχή της μη διάκρισης όλων των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην περιοριστεί στους πολίτες ορισμένων μόνο χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να εξετάσουμε την ε, κατάσταση των ενδοκινοτικών μεταναστών και να δούμε αν γίνονται σεβαστά τα δικαιώματά τους στις διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα επίσης ε, να, ε, να δώσουμε λίγη προσοχή και συγκατάσταση των Πολωνών πολιτών που ε, σε άλλες χώρες, μεταναστεύουν σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή ε, χωρών, ε, υπηκών τρι, άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταναστεύουν προς την Πολωνία. Κάθε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει δυνατότητα ελεύθερης διακίνησης και εγκατάστασης ε, στην επικράτη οποιασδήποτε χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προβλέπεται από τη συνθήκη. Και σίγουρα τα δικαιώματα αυτά θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Βέβαια, έχουμε μαζική αποδημία Πολωνών προ άλλε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Στι αρχέ του 2008, στι ευρωπαϊκέ χώρε, είχαμε περίπου 2 εκατομμύρια πολωνού, απόδημους Πολωνού. Κυρίω στην ε, ε, Μεγάλη Βρετανία, πάνω από μισό εκατομμύρια, περίπου μισό εκατομμύριο στη Γερμανία, 220.000 στην Ιρλανδία και 805.000 στην Ιταλία. Βέβαια, μια τέτοια μαζική έξοδος δείχνει τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Πολωνοί πολίτες ε, και εξηγεί ίσως τη μείωση της ανεργίας στην Πολωνία. Βέβαια, όλο και περισσότερο οι πολίτες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Ε, και υπήρξαν προβλήματα και με τους εργοδότες, ε, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομεί. Θα πρέπει επίσης να δούμε τις ε, περιπτώσεις που οι Πολωνοί δουλεύουν σε ενειδίκευτες θέσεις και δεν έχουν πάντα τη δυνατότητα να ασκούν τα δικαιώματα που έχουν οι πολίτες της χώρας υποδοχής. Υπάρχει μια φαιά ζώνη της οικονομίας και σε ακραίες περιπτώσεις οι Πολωνοί γίνονται θύματα σχεδόν δουλεμπορίου. Πολλοί Πολωνοί που βρίσκονται στην Αλοδαπή δεν ξέρουν ότι έχουν δικαίωμα σε μια αξιοπρεπή εργασία και δεν ασκούν όλα τους τα δικαιώματα. Δεν έχουν τα δικαιώματα, δεν ασκούν τα δικαιώματα απόκτησης και ε, κατάλληλης ποιοτικής παιδείας και φίτησης σε ξένη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα λάβουμε υπόψη. Γιατί από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι σήμερα η ανεργία στην Πολωνία έχει αυξηθεί κατά 1,2%. τον Ιανουάριο περνούσε το 10%. Αυτό δείχνει την δύσκολη οικονομική κατάσταση στην Πολωνία. Αυτό συνδέεται μερικές φορές και με την επιστροφή των Πολωνών από τις υπόλοιπες κοινοτικές χώρες όταν έχασαν τη θέση τους εκεί. Επίσης, έχουμε μετακίνηση των Πολωνών ενδοκινοτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετακινούνται από μια χώρα όπου έχασαν, τις, έχασαν την απασχόλησή τους σε μια άλλη χώρα που θεωρούν ότι θα αποκτήσουν αλλού καλύτερες, ικανό, δυνατότητες. Για παράδειγμα, από την Ισλανδία και την Μεγάλη Βρετανία πολλές φορές μετατοπίζονται προς την Ορβηγία. Οι Πολωνοί ελπίζονται ότι εκεί θα βρουν καλύτερες θέσεις απασχόλησης. Όλα αυτά χρειάστηκαν μια εντατικοποίηση των προσπαθειών της, του, του Πολωνικού Υπουργείου Εσωτερικών για τη διευκόλυνση της επιστροφής των Πολωνών. Το 2007 είχαμε μια, ε, τον ειδικό σύμβουλο και μάλιστα συστήθηκε ειδική επιτροπή για τη διευκόλυνση των θεμάτων επαναπατρισμού των Πολωνών. Η ομάδα αυτή εργασίας θα εκπονήσει ειδικό εγχειρίδιο και θα κατασκευάσει ειδική ιστοσελίδα για τους ε, απόδημους Πολωνούς που ενδιαφέρονται να επαναπατριστούν στην Πολωνία. Επίσης, προτάθηκαν κάποια μέτρα φορολογικής απαλλαγής για τους ε, απόδημου που θέλουν να επιστρέψουν στην Πολωνία, προκειμένου να ξεκινήσουν μια οικονομική δραστηριότητα. Σα παρέθεσα τη θέμα, την περίπτωση των Πολωνών που εργάζονται στην Αλοδαπή. Οι Πολωνοί έχουν αντίστοιχα προβλήματα με τους ε, μετανάστες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δουλεύουν στην Πολωνία που έχουν αντίστοιχα προβλήματα. Η Πολωνία γίνεται όλο και πιο σημαντικό οικονομικό εταίρο, βρίσκεται σε μια πολύ ελκυστική γεωρική θέση και έχει όλο και καλύτερα οργανωμένη υποδομή. Το 2008, 7.500 πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσαν διαμονή στην ε, Πολωνία. Περισσότεροι ήταν Γερμανοί και σε δεύτερη και τρίτη θέση έρχονταν οι Γάλλοι, οι Ιταλοί και κατόπιν οι Βούλγαροι. Όλο και περισσότεροι κοινοτικοί πολίτες θέλουν να εγκατασταθούν στην Πολωνία είχαμε, επαναλαμβάνω, πολίτες από τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία. Επίσης έχουμε πολίτες από, τρίτη, από τρίτες χώρες ε, στην Πολωνία. Για παράδειγμα, πολίτες της Ουκρανίας, ε, της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών κατέθεσαν ε, αιτήσει για απόκτηση της πολωνικής άδειας παραμονής στον περασμένο χρόνο. Όλα αυτά δείχνουν και μετά από δημοσκοπήσεις που κάναμε είχαμε πολύ ε, θετικές εντυπώσεις των Ευρωπαίων πολιτών για την ε, συμμετοχή της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλο και περισσότερους ε, Ευρωπαίους πολίτες έχουμε στην Πολωνία κάτι που καθιστά όλο και μεγαλύτερη την ανάγκη καλύτερης εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου και στην Πολωνία. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και, των τα δικαιώματα των οικογενειών τους είναι πολύ σημαντικό θέμα. Η Πολωνία υποστηρίζει αυτή την έκθεση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ για την εφαρμογή της οδηγίας και πιστεύω ότι θα πρέπει να βελτιωθεί από τα κρατημέλη ο τρόπος εφαρμογής αυτής της οδηγίας. Βέβαια υπάρχουν κάποια στοιχεία της οδηγίας που δημιουργούν ερμηνευτικά προβλήματα. Πιστεύω ότι όλα τα ερμηνευτικά αυτά προβλήματα θα αποσαφινιστούν με συζήτηση και αποκατάσταση διαφάνειας. Η καλύτερη, βελτίω, η καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας θα απαλλάξει πολλά, πολλά κράτη από τα προβλήματα. Χρειαζόμαστε όμως μεταβατικές διατάξεις. Θα πρέπει οι χώρες φιλοξενίας να βελτιώσουν τις διατάξεις ένταξης των μεταναστών στις κοινωνίες της. Επίσης έχουν παρατηρηθεί και πολλές καταχρήσεις στο δικαίωμα ελεύθερης διακίνησης. Έχουμε και τη σχετική νομολογία του ΔΕΚ. Για παράδειγμα την υπόθεση ΜΕΤΟΧ Το ΔΕΚ στην ομολογία του μας υπεθυμίζει ότι στα πλαίσια της οδηγίας 1308 του 2004 του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου τα θέματα δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών και των μελών της οικογένειάς τους που διακινούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση αυτά κάθε πολίτης Ένωση έχει δικαίωμα ε, διακίνησης και διαμονής σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να τύχει της ε, ασφάλειας υγείας χωρίς να επιβαρύνει το σύστημα κοινωνική ασφάλεια. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν δικαίωμα διακίνησης ε, με βάση την ηθαγένεια αυτή σε οποιοδήποτε κράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σύζυγος του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που διαμένει σε τρίτη χώρα και που συνοδεύει τον πολίτη αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να, να επωφεληθεί από τις διατάξεις οδηγής ανεξάρτητα από την ημερομηνία σύναψης ε, του γάμου και ανεξάρτητα από το πότε ε, έφυγε από το τρίτο κράτος. Σε ό,τι αφορά την ομολογία ΜΕΤΟΚ ε, και άλλων, πολλές φορές διαπιστώνονται καταχρήσεις στην εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την νομιμοποίηση της ε, διαμονής των μελών της οικογένειας. Βέβαια, το θέμα της ε, ελευθερομετανάστευσης είναι πολύ σημαντικό και απειλεί μερικές φορές ε, τις προσπάθειες του, του κράτους για την βελτίωση κατάστασης των νόμιμων μεταναστών. Επίσης, οι πολωνικές διατάξεις για το δικαίωμα διαμονής στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και της ε, διαμονής των μελών δεν έχουν προκαλέσει άσκηση προσφυγών μέχρι στιγμής. Οι πρόσφατες στρατηγικές μας δείχνουν ότι δεν υπάρχουν καταχρήσεις ε, ούτε το ούτε το 2008 στην Πολωνία σε σχέση με τα δικαιώματα αυτά, ούτε και εκδόθηκε καμία απόφαση για απόρριψη άδεια παραμονή ε, μέλους τη οικογένειας ε, μετανάστη που ζει στην Πολωνία. Επίση, θα ήθελα να τονίσω ότι η πολωνική κυβέρνηση υποστηρίζει την έννοια της ευρωπαϊκής Ιθαγένεια, γιατί κατά τη γνώμη μα, τα δικαιώματα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας είναι πολύ σημαντικά και χρειαζόμαστε φυσικά και στην εθνική μας οικονομία αλλοδαπούς επενδυτές και εργαζόμενους από άλλες χώρες μέλη. Η ελεύθερη διακίνηση των προσώπων είναι από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ενισχύουν την συμμετοχή της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σόρεν για μια εξαντλητική στην πληρότητα της παρουσίασης για τον τρόπο με τον οποίο οι πολωνικές αρχές αντιμετωπίζουν το θέμα της ελευθερίας διακίνησης και εγκατάστασης. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Γκαλίτσκι πρώτα, αλλά θα ήθελα να μάθω αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελα να πάρω το λόγο σε αυτή τη φάση. Δίνω λοιπόν το λόγο στον κύριο Γκαλίτσκι. Παρακαλώ όχι πάνω από πέντε λεπτά. Προσπαθώ να κερδίσω λίγο από το χρόνο τον οποίο έχουμε μέχρι τώρα σώρευση. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζοντας την ομιλία του κυρίου Διευθυντού, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή μας στις τεράστιες προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα των φορέων που ασχολούνται με τα προβλήματα και τις προαπτικές της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Όπως είπε και ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κυβέρνησης, ο κ. Μπαρό, ο Ευρωπαϊκό, Ευρωπαίος πολίτης δεν είναι μια, ένα φανταστικό μόρφωμα. Έχει γίνει πια μια απτή πραγματικότητα. Έχει γίνει ένας Ευρωπαίος πολίτης που χαίρει συγκεκριμένων δικαιωμάτων αλλά φέρει και αντίστοιχε υποχρεώσεις. Και κυρίως ε, ε, έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις απέναντι στην Ένωση καταρχήν, απέναντι στην ε, πατρίδα του, αλλά και απέναντι σε τρίτες, στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε η νομική θέση του Ευρωπαίου πολίτη οριοθετείται και με βάση τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχει απέναντι σε αυτού του τρει φορεί, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την πατρίδα του και τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έκθεση κυρίας Γκάτσεκ μιλάει για ανάγκη ενίσχυσης των δικαιωμάτων του πολίτη που απορρέουν από, δικαιωμάτων του πολίτη που απορρέουν από την ιδιότητα της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Για παράδειγμα, θα πρέπει να ενισχύσουμε την διπλωματική και προξενική προστασία. Αυτή τη στιγμή, ας είμαστε ειλικρινείς και μάλιστα υπό το φως των πρόσφατων περιστατικών που είχαμε στη Βομβάη, διαπιστώνουμε ότι το θέμα της διπλωματικής και προξενικής προστασίας πόρα απέχει από, την επιθυμητή, από τον επιθυμητό στόχο. Επίσης, θα πρέπει να δούμε το θέμα της ε, μετανάστευσης, ε, της εσωτερικής μετανάστευσης και της προστασίας των ε, μεταναστών και των μελών της οικογένειάς τους και την ίση, ίση μεταχείρισή τους με τους πολίτες της χώρας φιλοξενίας. Θα πρέπει να σκεφτούμε και το θέμα των νέων δικαιωμάτων στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Ιδιαίτερα μετά την δεχόμενη θέση σε ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας. Νομίζω ότι μετά την θέση σε ισχύ της ηθίκης της Λισαβόνας θα μπορούσαμε να διευρύνουμε αυτό το κατάλογο, να διευρύνουμε αυτό το κατάλογο με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Η ιδέα της ευρωπαϊκής ηθαγένειας θα πρέπει να περάσει από το ιδεολογικό επίπεδο το συντομότερο δυνατό στην πράξη, να μετατραπεί σε ένα νομικό καθεστώς που γεννά συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Συνθήκη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τα δικαιώματα που αναγνωρίζει εκεί. Επίσης έχουμε το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων. Εκεί έχουμε έναν ολόκληρο κατάλογο με νομικά δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Πραγματοποιώντας λοιπόν όλα αυτά τα δικαιώματα θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση ώστε ένα από τα θεμελιώδη δικαιώματα στους, του Ευρωπαίου πολίτη να είναι για αυτό τη ελεύθερης διακίνησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Γκαλίτσκι. Θέλει κάποιος άλλος το λόγο σε αυτή τη φάση. Ο Παναγιώτης. Ε, volontaire ou moralement contraint ναι. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, θα είμαι σύντομος και θα πω ε, κάτι σε επέκταση των όσων έχουν λεχθεί και από τον κύριο Μπαρό και από την κυρία Ούρσουλα Κάτε. Τα δικαιώματα είναι εκεί. Τα άρθρα 17 ως 20 της Συνθήκης Ευρωπαϊκής Κοινότητας καθορίζουν τα δικαιώματα αυτά όπως και άλλα πρόνοια στο συνθήκο. Ένα σημείο θέλω να δείξω. Τα ξέρουν αυτά οι πολίτες της Ευρώπης και αν δεν τα ξέρουν γιατί δεν τα γνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά. Και αν τα γνωρίζουν πόσο ωφέλιμα είναι σε αυτούς και πόσο τα χρειάζονται αυτά για να νιώθουν μια διασύνδεση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι τα ερωτήματα που πρέπει να απασχολήσουν και εμάς και όλους εκείνους οι οποίοι ενδιαφέρονται να προωθήσουν την ευρωπαϊκή ιδέα γιατί φιλολογούμε κάποιοι που είμαστε περίπου το ελίτ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε είναι πολιτικοί, είτε είμαστε ε, ηγετικοί παράγοντες, αλλά προχωρούμε εμείς μόνοι μας και οι πολίτες μένουν πίσω και δεν τους συνδέομαι με αυτά που μας απασχολούν εμάς. Και εδώ είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γι' αυτό και στις τροπολογίες που θα καταθέσω στην έκθεση της Ούρσουλα και σε αυτή την έκθεση που είχα καταθέσει εκ μέρους τη συνταγματικής, της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων θίγω ακριβώς αυτό το θέμα. Ότι η Επιτροπή και όλοι μας πρέπει να κάνουμε προγράμματα πολιτικής αγωγής του Ευρωπαίου πολίτη. Να ξέρει τα δικαιώματά του και να τα χρησιμοποιεί ταυτόχρονα. Να τα εκτιμήσει. Όχι να τα ξέρει απλώς θεωρητικά. Και καταλήγω κύριε Πρόεδρε με το να πω ότι το Κοινοβούλιο έχει δύο εκθέσεις αυτή τη στιγμή. Έχουμε την έκθεση της κυρίας Βάλεαν που απασχολείται με το δικαίωμα εγκατάστασης και διακίνησης των Ευρωπαίων πολιτών, που είναι πολύ βασική έκθεση. Έχουμε και την έκθεση της κυρίας Γκάτζεκ. Και οι δύο εκθέσεις θα περάσουν, θα προωθηθούν, θα φιλολογήσουμε και πάλι θα πούμε τα δικαιώματα, αλλά δεν αγγίζουμε και τα ουσιαστικά προβλήματα. Γιατί ο τίτλος των εκθέσεων μας είναι προβλήματα και προοπτικές. Και δεν φταίμε εμείς. Φταίει και η, πρώτη, η πέμπτη έκθεση της Επιτροπής, η οποία αντί να μας πει για τα προβλήματα, μας απαριθμεί τα δικαιώματα που ξέρουν. Εμείς τουλάχιστον. Γι' αυτό πρέπει να αγγίξουμε το πρόβλημα. Και το πρόβλημα ποιο είναι. Ποια είναι τα προβλήματα και οι προοπτικές και τι είναι που πρέπει να ξέρουν και πώς τα ε, σχέση με τα δικαιώματα του πολίτε και πώς να ασκήσουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Ευχαριστώ Παναγιώτη. Νομίζω ότι οι επόμενοι ομιλητές θα έχουν την δυνατότητα να δώσουν κάποιες απαντήσεις στα ερωτηματικά που έθεσες και η Ούρσουλα επίσης με τη σειρά της θα επανέλθει σε κάποια από αυτά τα στοιχεία στα συμπεράσματά της. Δίνω το λόγο λοιπόν στον δεύτερο μιλητή για σήμερα το απόγευμα, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή, τον κύριο Διαμαντούρο. Ο κύριος Διαμαντούρος ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι προσδοκίες των πολιτών από τα ευρωπαϊκά όργανα. Συσταγωγικά θα έλεγα πληρώνεται γι' αυτό και πρέπει να μας πει ποια είναι η δυσφορία και δυσθυμία που νιώθει ο Ευρωπαίος πολίτης. Του δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Άκουσα τις παρατηρήσεις του κυρίου Δημητρίου με προσοχή. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα πλαίσια της απάντησής μου για τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις σχέσεις ανάμεσα στα ευρωπαϊκά όργανα και τον πολίτη. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, λέει ο κ. Διαμαντούρος που μιλούσε μέχρι τώρα γαλλικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να πάρω μέρος σε αυτή την ακρόαση. Χαίρομαι που έχω την δυνατότητα να μοιραστούμε απόψεις για την ανάπτυξη της ιδιότητας και της ευρωπαϊκής ηθαγένειας μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω μια καλή πρώτη εικόνα για το τι πιστεύει ο Ευρωπαίος πολίτης και η κοινωνία των πολιτών και από τα γράμματα που λαμβάνω και από τις επαφές μου σε ταξίδια. Αυτά με κάνουν να πιστέψω ότι οι Ευρωπαίοι εκτιμούν και αξιολογούν θετικά πολλές πλευρές των ευρωπαϊκών νομικών ρυθμίσεων, το δικαίωμα μετακίνησης, το δικαίωμα ισότητας αντιμετώπισης. Υπάρχουν και άλλα δικαιώματα κάποιων κατηγοριών συγκεκριμένων πολιτών όπως ε, οι ταξιδιώτες με αεροσκάφη κτλ. Το πρόβλημα για πολλούς Ευρωπαίους είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά διοικητικά εμπόδια και αυτά τα εμπόδια κάνουν δύσκολα να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν σωστά τα δικαιώματα τα οποία έχουν. Υπάρχουν θέματα για την διαφάνεια, υπάρχουν θέματα για την έλλειψη της διαφάνειας και τα περισσότερες, οι περισσότερες αναφορές που έρχονται σε μένα και τα παράπονα αφορούν τα ευρωπαϊκά όργανα και είναι λογικό γιατί εγώ με αυτά ασχολούμαι. Αφορούν λοιπόν την διαφάνεια στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα σε θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο ισχύει και για τις επαφές των πολιτών, τις ανησυχίες μάλλον των πολιτών για τα επίπεδα δεοντολογίας σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και σε όργανα των κρατών μελών. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι υπάρχει μια δεδομένη αντίληψη για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια που βασίζεται στα δικαιώματα, στην σωστή χρήση και σεβασμό των δικαιωμάτων και στην πολιτική δεοντολογία. Θα αναφερθώ αναλυτικότερα σε αυτά τα στοιχεία. Να θυμίσω όμως πρώτα πως η ευρωπαϊκή ηθαγένεια συμπληρώνει την εθνική ηθαγένεια και δεν την αντικαθιστά αντικατοπτρίζει την διτή φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών. Κάθε κράτος μέλος έχει το δικό του σύνταγμα, τα δικά του πολιτικά όργανα, ταυτόχρονα όμως είναι σημαντικός πρωταγωνιστής στο θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης. Γι' αυτό τον λόγο δεν θα πρέπει να συζητάμε μόνο απομονωμένα τις σχέσεις του πολίτη ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και τις σχέσεις του πολίτη με τα εθνικά όργανα για τα ευρωπαϊκά θέματα και τα ευρωπαϊκά πράγματα. Απαιτείται φυσικά κατά πρώτον η χρηστή διαχείριση των δικαιωμάτων των πολιτών. Δεν έχουμε χρόνο για να αναλύσουμε την έννοια της χρηστής διαχείρισης. Θα ήθελα δύο θέματα να υπογραμμίσω. Πρώτον, θα πρέπει οι νομικές ευρωπαϊκές ρυθμίσεις να λειτουργήσουν αποτελεσματικά. Δεν θα πρέπει μόνο να εφαρμόζουμε τους νόμους. Αν δεν εφαρμόζονται σωστά και δεν επιβάλλονται σωστά... Αλλιώς δεν θα έχουν καλά αποτελέσματα. Δεύτερον, που έχει σχέση με το πρώτο σαφώς, οι πολίτες θα πρέπει να έχουν διαθέσιμα ένδικα μέσα αποτελεσματικά αν τα δικαιώματά τους δεν γίνουν σεβαστά η ευθύνη για την εφαρμογή του δικαίου είναι των κρατών μελών. Γι' αυτό πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό δίκαιο μπορεί να είναι αποτελεσματικό μόνο αν μπορέσουμε να προωθήσουμε μία έννοια ιδιοκτησίας μεταξύ των δημοσίων διοικήσεων των κρατών μελών. Αν ε, το θεωρούν κάτι εξωτερικό που τους επιβάλλεται από τις Βρυξέλλες, ε, το ευρωπαϊκό δίκαιο και όχι ένα σώμα που περιέχει κανόνες που λαμβάνουν υπόψη ευαισθησίες και ιδιαιτερότητες, τότε δεν θα υπάρχει η προθυμία να εφαρμόζεται πλήρως. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών προάγει την καλή εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Δικαίου σε επίπεδο κρατών μελών και αποτελεσματικά ενδικά μέσα οι συνάδελφοι ε, λαμβάνουν υπόψη και τα θεμέλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει επίσης να εφαρμόζεται με τρόπο δίκαιο αποτελεσματικό ε, από τις αρχές των κρατών μελών. Η κοινότητα των διαμεσολαβητών στην Ευρώπη δεν μπορεί όμως από μόνη της να κάνει το ε, έντονο lifting που χρειάζεται σε εθνικό επίπεδο. Για να υπάρχει αίσθηση ιδιοκτησία τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τα Ευρωπαϊκά Κοινοβούλια πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στι νομοθετικέ διαδικασίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πράγμα που προβλέπει η συνθήκη τη Λισαβόνα. Πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο στην παρακολούθηση τη εφαρμογή τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και θα πρέπει να λογοδοτούν οι δημόσιες αρχές για οποιασδήποτε ελλείψεις. Αν περάσουμε τώρα στο θέμα της διαφάνειας, ε, σημαντική πρόοδος επετέχθη σε επίπεδο θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κανονισμός για την ασφάλεια, ο κανονισμός 149 του 2001 δηλαδή, εφαρμο... Ε, ε, αφορά την πολιτική πριν από την νομοθεσία, την νομοθετική διαδικασία και την λειτουργία των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων μετά τη θέσπιση των ευρωπαϊκών κανόνων. Για παράδειγμα, η Κομισιόν δημοσιεύει την ανάλυση αντικτύπου, επιπτώσεων, πολιτικών προτάσεων ε, και με βάση τις εκτιμήσεις του Συμβουλίου ή του Φορέα Αξιολόγησης επίσης προβλέπεται και θεσμοθετημένος ρόλος των λόμπι. Αυτό ε, προάγει την διαφάνεια παρόλο που υπάρχει ακόμη περιθώριο για πολλές περισσότερες βελτιώσεις. Ό,τι αφορά την νομοθετική διαδικασία τον Οκτώβριο του 2005 συνέστησα το Συμβούλιο να συνεδριάζει δημοσία όποτε συζητεί νομοθετικά θέματα. Το 2006 η Ευρωπαϊκή ε, Επιτροπή υιοθέτησε ένα ε, ψήφισμα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Συμβούλιο όμως ακόμη δεν συμμορφούται απόλυτα με τη σχετική σύσταση. Η πλήρης διαφάνεια της νομοθετικής διαδικασίας στο Συμβούλιο ενισχύει την υπηκότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι Ευρωπαίοι μπορούν να παρακολουθούν τι κάνουν ε, οι κυβερνήσεις τους που έχουν εκλέξει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολίτες της Ένωσης μπορούν να παρακολουθούν αποτελεσματικότερα το έργο ενός ζωτικού θεσμικού ε, οργάνου. Επίσης ε, έχουν γίνει και σε εθνικό επίπεδο πρόοδοι για την διαφάνεια δικαιούχοι χρηματοδότησης ευρωπαϊκής. Γενικότερα οι πολίτες που θέλουν να γνωρίζουν πώς εφαρμόζονται οι ευρωπαϊκοί νόμοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διαπραγματεύονται, αν θέλετε, με 24, 24, σετ κανόνων. Ε, δηλαδή να λάβουν υπόψη και τα 27 εθνικά νομικά πλαίσια. Για να αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες για διαφάνεια θεωρώ ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μοιράζονται πληροφορίες και ευέλτιστες πρακτικές για, ε, με πρόσβαση στην ενημέρωση και στα ευρωπαϊκά έγγραφα. Είμαι πρόθυμος να εργαστώ με τους εθνικούς επιτρόπους ε, σε, θέματα πληροφόρησης ούτως ώστε να συμβάλλουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση. Περνώ στο τρίτο στοιχείο της αντίληψης της υπηκότητας ε, δεοντολογία στη δημόσια ζωή. Τα πρότυπα σε αυτό το τομέα διοντολογίας είναι απαραίτητα διότι συμβάλλουν στην ε, συνειδητοποίηση της λογοδοσίας και της ε, εμπιστοσύνης. Δεν θα επανεφεύρω με τον τροχό. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης, πολλά κράτη-μέλη, διεθνείς οργανισμοί όπως όσα ε, έχουν όλοι κάνει πολύτιμο έργο στον τομέα της δεοντολογίας στο δημόσιο. Όπως όμω και με τα θέματα δημόσια διοίκηση και της διαφάνειας, οι προσδοκίε των πολιτών δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με, τεχνική, με τον τεχνικό διαχωρισμό μεταξύ θεσμικών οργάνων Ευρωπαϊκή Ένωση και κρατών μελών από την άλλη. Αυτό που χρειάζεται θεωρώ είναι οι πολίτες με, ε, διακριτό και σαφή τρόπο να ε, ισχύουν οι αρχές που αφορούν και τις, ε, τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα αλλά και τους κανόνες λειτουργίας των εθνικών αρχών. Οι αρχές δεν πρέπει να θεωρηθούν ότι επιβάλλονται από τις Βρυξέλλες αλλά ότι είναι η απόσταξη των βέλτιστων πρακτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα. Όταν, συναντώ, όταν θα συναντήσω τους εθνικούς διαμεσολαβητές στην ε, διετή διάσκεψη θα συζητήσουμε αν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάποιες αρχές δεοντολογίας ως περαιτέρω συμβολή από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διαμεσολαβητών ώστε η υπηκότητα στην Ευρώπη να γίνει μια ζώσα πραγματικότητα. Συμπεραίνοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι η υπηκότητα είναι μια ηθαγένεια είναι ε, μια ε, έννοια που περιλαμβάνει μεγάλο πλούτο είναι ένα μέσο να αποκτήσουν ε, δυνατότητες όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι Ευρωπαίοι πολίτες, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Η εστίαση αντικατοπτρίζει τις συγκεκριμένες ε, ανησυχίες που έχουν ε, να εκφράσουν σε μένος διαμεσολαβητή. Επίσης, το, ένα τέτοιο κοινοβούλιο θα πρέπει ε, μια τέτοια προσπάθεια θα πρέπει να είναι πολιτική προτεραιότητα γιατί το, θα πρέπει, η ηθαγένεια σημαίνει ε, ότι ανήκουμε σε μια ευρεία κοινότητα με υποχρεώσεις, δικαιώματα, ε, λογοδοσία, δυνατότητα συμμετοχής στα κοινά. Η ανάπτυξη της έννοιας της ηθαγένειας αφορά την ποιότητα της δημοκρατίας. Ενισχύει την νομιμότητα των ε, πολιτικών ε, θεσμικών οργάνων. Ιδιαίτερα ε, στα πλαίσια της παρούσας οικονομικής κρίσης θα πρέπει να τονίσουμε ότι η νομιμότητα είναι πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο σε όλους μπορεί να αποφέρει ωφέλη. Αν συνεργαστούμε με διαφάνεια, με διοντολογία τα, τα διαφανή θεσμικά όργα ε, αποκτήσουν νομιμότητα στα μάτια των πολιτών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, Ευχαριστώ κύριε Διαμαντούρο για την παρουσίασή σας. Δίνω το λόγο τώρα στους υπόλοιπους συναδέλφους οι οποίοι θα ήθελαν το λόγο να θέσουν μια συμπληρωματική ερώτηση να εκφράσουν μια κριτική ή να πούνε ένα καλό λόγο. Ούτε τόνα ούτε τ' άλλο, σας έπεισαν όλοι, μας πείσατε μάλλον. Ευχαριστώ λοιπόν και τον κύριο Διαμαντούρο. Δίνω... Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Θα δώσουμε το λόγο στον Ερνέστο Μπιάνκι ο οποίος είναι υπεύθυνος για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα θεμελιώδη δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μας μεταφέρει τη γραφειοκρατική αντίληψη για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να σας συγχαρώ για αυτή την πρωτοβουλία Πράγματι οι απόψεις μου θα είναι κάποιες απόψεις γραφειοκρατών, αλλά όχι μόνο. Έχουμε πάρα πολλές επαφές με τους πολίτες, οι οποίοι φαίνεται ότι γνωρίζουν ποια είναι τα δικαιώματά τους και μας το θυμίζουν αυτό όταν έρχονται σε εμά και ζητούν ε, αρρωγή. Βέβαια αυτό είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτών με τους οποίους έρχεται σε επαφή ο κύριος Διαμαντούρος θα ήθελα να υποστηρίξω όλα όσα είπε ο κύριος Διαμαντούρος άλλωστε. Είναι δύσκολο όταν έρχεται κανείς σε ατομικά προβλήματα να ασχολείται με αυτά από τις Βρυξέλλες. Είμαστε ίσως μερικές φορές πολύ μακριά και το ότι η τοπική, εθνική διοίκηση μερικές φορές δεν γνωρίζει ορισμένες από τις δυνατότητες τις οποίες έχουμε, αυτό είναι αλήθεια. Γιατί υπάρχουν πάντα ορισμένοι κανόνες οι οποίοι ναι μεν φαίνονται απλοί όταν τους διαβάζει κανείς σε μια πρώτη φάση, αλλά παρόλα αυτά αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο από υπηρεσίες που μπορεί να απέχουν η μία από την άλλη μόνο 20 χιλιόμετρα και αυτό δημιουργεί ένα πολύ μεγάλο αριθμό παραπώνων και ανεξάρτητα από το πόσο μπορεί κανείς να εμπλουτίσει το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν μπορεί κανείς να τα διαχειριστεί όλα από τις Βρυξέλλες. Θα πρέπει λοιπόν τα δικαιώματα των πολιτών όπως υπάρχουν στις συνθήκες σήμερα να εφαρμόζονται αποτελεσματικά Υπάρχουν δύο τομείς στους οποίους θα πρέπει κάτι να κάνουμε και αυτό θα φανεί ή φαίνεται μάλλον και στην έκθεση την οποία παρουσιάσαμε συνοδευτική της 2048 επικοινωνία και εφαρμογή. Σε επίπεδο επικοινωνίας πρέπει να πάμε καλύτερα, όχι μόνο στις επαφές μας με τους μεμονωμένους πολίτες, αλλά να πάμε καλύτερα και στις επαφές μας με τις τοπικές αρχές. Προετοιμάζουμε κατευθυντήριες γραμμές οι οποίες θα βοηθούν τα τοπικά επίπεδα εξουσίας να εφαρμόζουν την οδηγία 2004-48. Πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα εθνικό συμπλήρωμα στις απλουστευμένες κατευθυντήριες γραμμές και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε με πιο σωστό τρόπο τους νόμους αυτούς. Για την εφαρμογή έχουμε πολλά να κάνουμε με τα κράτη-μέλη. Είμαστε τώρα σε μια διαδικασία ε, συζήτησης όλων των δύσκολων θεμάτων. Ε, ε, τα δύσκολα θέματα που προέκυψαν σε σχέση με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας που είναι κέρια σημασία, η 238, για την ηθαγένεια και πρώτα απ' όλα προσπαθούμε μαζί με τις εθνικές ορχές να καταλήξουμε στις δυσκολίες όπως τις βλέπουν εκείνες. Η προβληματική εφαρμογή αποτελεί πρόβλημα πολλές φορές επίσης ε, καμιά φορά Υπάρχουν, ε, ε, ε, είναι πιο εύκολο να δει κανεί ε, προβλήματα σε σχέση με νομοθεσία από το Εθνικό Κοινοβούλιο. Μπορεί να υπάρχει κάποιος κανονισμός από κάποια κοινότητα σε μικρό επίπεδο τοπικό επίπεδο και δεν αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα μέχρι ότου μας επιστήσει κάποιος την προσοχή. Πρέπει λοιπόν εδώ να εργαστούμε περισσότερο και με τα Εθνικά Κοινοβούλια ακόμη, ούτω ώστε ε, και αυτό θα μπορούσε να το κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κάνει υποθέτω για να φροντίσει ώστε τα εθνικά κοινοβούλια να ε, μας βοηθούν να παρακολουθούμε ε, τι συμβαίνει σε εθνικό επίπεδο στα κράτη-μέλη. Επίσης είδαμε και αποτυχίες σε σχέση με την προξενική προστασία. Η προξενική προστασία είναι ένας τομέας όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, εύχεται για το καλύτερο. Ελπίζομαι να μπορέσει να ακυρωθεί η συνθήκη της Λισαβόνας. Αν συμβεί αυτό θα υπάρχει για πρώτη φορά η ευκαιρία να θέσουμε επιτάπητος νομοθετικές προτάσεις ώστε να δώσουμε σάρκα και οστά στα δικαιώματα αυτά. Γιατί όντως είναι από τα πιο σύνθετα δικαιώματα δύσκολα ε, και πραγματικά σε σχέση με τη 238 μας αφορά όλους. Ε, δεν έχει σημασία αν μετακινηθήκαμε από το ένα κράτος μέλος στο άλλο μόνο. Επίσης, ε, έχουμε εδώ καταρτήσει ένα πρόγραμμα δράσης που ακούγεται γραφειοκρατικό, αλλά αντιμετωπίζουμε τεράστιες αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη ε, πάνω σε αυτό το θέμα. Πρώτον, γιατί ε, δεν είναι πρωτόγονοι σε ό,τι αφορά τα πρότυπά τους, έχουν πρότυπα, αλλά υπάρχουν πολλοί και διάφοροι κανόνες για την παροχή της προξενικής προστασίας. Είναι συνταγματικό δικαίωμα στη Δανία, αλλά ε, είναι μόνο ε, θέμα ε, ευγενούς προσφοράς στο Ηνωμένο Βασίλειο και αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα όχι μόνο σε περιόδους μεγάλων κρίσεων όπου το θέμα είναι οι μεγάλες δαπάνες και ποιος θα τις πληρώσει αλλά και σε ατομικό επίπεδο στο διεθνές δίκαιο υπάρχουν πολλοί κανόνες και διαφορές πολύ λεπτές μεταξύ της προξενικής υποστήριξης, επικούρησης ή προστασίας ή το ε, δικαίωμα που προβλέπει εξουσιοδότηση των προξενικών αρχών ε, της χώρας ε, από την οποία προέρχεται ο, ο, πολίτης που έχει πρόβλημα. Χρειάζονται απλουστεύσεις αν μπορούμε σε, πολλά, σε πολλούς τομείς λαμβάνοντας υπόψη και το ε, την προσθήκη του κειμένου του άρθρου 20 ε, που αφορά τα διαβατήρια και την προσθήκη του δικαιώματος αυτού εκεί. Για τις ευρω... Ε, ευρωεκλογέ, ο Αντιπρόεδρος Μπαρό ανέφερε ότι πρέπει να μάθουμε περισσότερα για τον λόγο της χαμηλής συμμετοχής στις ευρωεκλογέ όταν η υπήκοοι δεν είναι στην χώρα καταγωγής τους. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να διοργανώσουμε μια έρευνα μετά από αυτές τις εκλογές και θα ρωτήσω με πολύ συγκεκριμένα τους πολίτες ποιες δυσκολίες αντιμετώπισαν, αν υπήρξαν δυσκολίες ή μήπως δεν ήθελαν να συμμετάσχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές εκτός της ε, χώρας καταγωγής τους, πρώτον γιατί δεν μιλούν τη γλώσσα καλά, δεύτερον δεν γνωρίζουν τους πολιτικούς, γάμο για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Νομίζω ότι όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε για να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και σε αυτό το μέτωπο. Μια τελευταία παρατήρηση και σταματώ γιατί εγώ ήρθα εδώ για να ακούσω και όχι να μιλήσω τόσο. Η αντίστροφη διάκριση ε, όλο και περισσότερο μας προβληματίζει σύν το χρόνο. Υπάρχουν τάσεις σε κάποια κράτη-μέλη και η οικονομική κρίση μπορεί να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο τα πράγματα όπου είναι περίπλοκο για μένα να εξηγήσω σε μια κυβέρνηση ή σε έναν πολίτη γιατί η ευρωπαϊκή νομοθεσία παρέχει περισσότερα δικαιώματα από το εθνικό δίκαιο καμιά φορά. Το γεγονός ότι έχει ασκηθεί το δικαίωμα της ελεύθερης διακίνησης σημαίνει περισσότερα δικαιώματα για έναν Ιταλό ε, στην περίπτωση της διακίνησης από την περίπτωση όπου δεν υπήρξε ε, ε, διακίνηση, δηλαδή στην περίπτωση όπου δεν έφυγε από την Ιταλία. Δηλαδή ε, αναφέρθηκε αυτό ως μπόνους. Ε, ε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο μπόνους στο ευρωπαϊκό δικαίωμα και η ευρωπαϊκή ηθαγένεια και η εθνική ηθαγένεια εκεί έρχονται σε κάποια αντιπαράθεση μπορεί να τη τη συζήτηση. Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για, την για το εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης που είδα και μας παρουσίασε. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς, εμείς μας θυμήσατε το καλό πρόσωπο της Ευρωπαϊκής Γραφειοκρατίας. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θα ήθελε το λόγο για να συμπληρώσει ίσως αυτά που ακούσαμε. Η Ούρσουλα. Μία ερώτηση, όχι μόνο γιατί ήταν ευγενή στα σχόλιά του ο κύριος Μπιάνκη, τι ακριβώς είναι αυτή η αντίστροφη διάκριση. Είπατε ότι σαν Ιταλός που μετακινείται πολλές φορές θεωρείτε ότι έχετε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με το αν μένατε στην Ιταλία. Μπορείτε να μου δώσετε ένα παράδειγμα. Μια ιδέα ακούγεται ενδιαφέρουσα. πρέπει να δούμε τι μπόνους προσφέρουν, τι πλεονεκτήματα προσφέρει η κινητικότητα στον Ευρωπαίο πολίτη. Ένα παράδειγμα, θεωρητικό βέβαια λίγο, η ύπαρξη αντίστροφης διάκρισης έχει σχέση με τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζουν το κοινοτικό δίκαιο τα κράτη-μέλη. Συνδέεται επίσης με την κατάσταση των πραγμάτων εφαρμογής της εθνικής νομοθεσίας στον ίδιο τομέα. Στη Δανία, σαν παράδειγμα σήμερα, και θα σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, αν θέλετε να παντρευτείτε κάποιον από μια τρίτη χώρα, αν τον παντρευτείτε αυτόν στην Δανία και είστε Δανός και δεν έχετε φύγει ποτέ από τη Δανία, οι κανόνες της Δανίας θα εφαρμοστούν. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορείτε να παντρευτείτε το συγκεκριμένο πρόσωπο εάν είναι παράνομος μετανάστης, αν έχει μητρό, αν έχει υπάρξει δηλαδή παράνομος μετανάστης σε άλλο χώρο ή αν δεν έχει αρκετούς πόρους για να επιβιώσει μέχρι τη στιγμή που θα παντρευτεί. Όλα αυτά δεν ισχύουν αν είστε ένας Ιταλός που πηγαίνετε στη Δανία σύμφωνα με τον κοινοτικό νόμο να εγκατασταθείτε ή αν σαν Δανός έχετε ζήσει σε μια άλλη χώρα έχετε χρησιμοποιήσει τον κοινοτικό νόμο και επιστρέφετε είτε με τον την σύζυγο ή ο τον τη σύζυγος σας σε επισκέπτεται εκ των υστέρων. Υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Ευχαριστώ. Δεν παρέλειψε κανέναν, ζήτησε κανείς το λόγο και δεν τον έλαβε. Να μην έχουμε διαμαρτυρίες μετά. Σας ευχαριστώ κύριε Βιάνκη και θα δώσω το λόγο στον επόμενο μας ομιλητή που από ό,τι βλέπω θα μας μιλήσει για τις προτεραιότητες και τις μελλοντικές εργασίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Το λόγο έχει ο κύριος Τόνι Βέναμπλς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θέλετε Venable, θέλετε Venables. Χαίρομαι ιδιαίτερος που βρίσκομαι στην δημόσια ακρόαση. Έπρεπε κανονικά να είμαι στη Βαρσοβία. Ε, low income. Σε μια διάσκεψη για μετανάστες χαμηλού εισοδήματο που αντιμετωπίζουν προβλήματα σε άλλες α, ε, ε, χώρες μέλη σε συνεργασία με τον α, Πολωνό διαμεσολαβητή. Και θυμήθηκα ότι είναι πολύ πιο εύκολο να κανεί Ευρωπαίο πολίτη, αν είναι καλά ενημερωμένο για τα δικαιώματά του, αν είναι μορφωμένο και αν έχει φυσικά δουλειά. Αλλά η Λιδία ε, ε, βρίσκεται όταν κάποιος ασχολείται με ενδοκινοτικούς μετανάστες που αντιμετωπίζουν όμως ε, δυσκολίες. Κάτι που δεν αναφέρθηκε ακόμη εδώ είναι ότι σε τελική ανάλυση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο μας δείχνει την ακολουθητέα πορεία. Και έχουμε βρεθεί εγκλωβισμένοι μεταξύ των προβλημάτων και των προοπτικών της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας γιατί το ΔΕΚ υιοθέτησε ένα μια συμβολική ερμηνεία για τη συνθήκη του, Μα, Μάστριχτ και με την ομολογία του σε 30 και πάνω αποφάσει, έδωσε στου ε, Ευρωπαίους πολίτες ε, περισσότερα δικαιώματα αυτά που νόμιζαν ότι είχαν. Οι μετανάστες στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να δικαιολογήσουν την ε, ελεύθερη διακίνησή τους ως θεμελιώδης δικαίωμα. Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να δικαιολογήσουν οποιοδήποτε περιορισμούς που εφαρμόζουν ως ε, αναλογικούς και ορθολογικούς. Γιατί βέβαια η ελεύθερη διακίνηση δεν ε, ισχύει ανεφόρων, αλλά δεν θα πρέπει όλοι αυτοί να συνδέονται με, με το οικονομικό επίπεδο του μετανάστη. Και ευτυχώς το ΔΕΚ γίνεται όλο και πιο κοινωνικό από αυτή την άποψη στην ε, νομολογία του. Το γραφείο μας έχει πάνω από 10.000 ε, αναφορές κάθε χρόνο ε, προσφυγές που εξετάζει από πολίτες. Και αυτό που μας ε, προβληματίζει είναι γιατί τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για να αναπτύξουν αυτή την ιδέα της ηθαγένειας της Ένωσης. Ενώ η νομολογία του ΔΕΚ είναι αρκετά πρωτοπόρα αυτό και συνήθως όταν προχωρεί το ΔΕΚ ακολουθούν τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα. Γιατί όμως δεν υπάρχει αυτή η πρωτοβουλία. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή αδιαφορία για το θέμα της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και όταν ολοκληρωθεί η δημόσια αυτή ακρόαση όλοι θα επιστρέψουμε σε πιο απτά θέματα. Και αν ρίξετε μια ματιά στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα διαπιστώσετε ότι η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι μια ε, σφαιρική έννοια αλλά έχει μείνει εδώ και πολλά χρόνια. Είμαστε ακόμη στην τέταρτη έκθεση και όχι ε, στην πέμπτη έκθεση. Και όταν ε, αποστέλλεται μία αναφορά στην, ε, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με θέμα την Ευρωπαϊκή Θεγενία, μας παραπέμπουν στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων, κάτι που δεν ήταν το ζητούμενο στην αναφορά μας. Φαίνεται ότι υπάρχει αρκετή αντίσταση και από πλευρά εθνικών κυβερνήσεων και η κατάργηση των συμβόλων της Ένωσης από την Συνταγματική Συνθήκη το κατέδειξε. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο ε, εφαρμόζεται η οδηγία για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια πόρο απέχει από την ομολογία και το πνεύμα του ΔΕΚ. Εφαρμόζεται μέσω μεταναστευτικών πολιτικών, μέσω πράξεων για αλλοδαπούς, μέσω, για, μέσω νομοθεσίας για αλλοδαπούς ή μετανάστες δεν περνάει το μήνυμα της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας στα κράτη-μέλη, ώστε να εφαρμόσουν όχι μόνο τον τύπο, αλλά και το πνεύμα του νόμου, όχι μόνο το γράμμα. Έχω τέσσερις συστάσεις για το μέλλον, τις μελλοντικές προτεραιότητες. Η έκθεση που εξετάζεται και αποτελεί τη βάση της δικής της έκθεσης, η πέμπτη έκθεση λοιπόν για την ηθαγένεια της Ένωσης, θα πρέπει να γίνει πιο ουσιαστική μέχρι ό,τι εκπονηθεί και η έκτη έκθεση. Θα πρέπει να βρεθεί στο επίκεντρο της συζήτησης σε συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Γιατί όπως είπε και ο Επίτροπος Μπαρό, είναι αυτή είναι αρκετά κατακαιρματισμένη και χρειαζόμαστε ένα είδος γενικού επιτελείου για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Θα πρέπει να φέρουμε στην Τράπεζα των Διαπραγματεύσεων ε, φορεί διαφορετικών αντιλήψεων και προοπτικών για την Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Και από τον ε, Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή ζητήσαμε κάποια εχέγγυα, κάποιες Την επόμενη φορά που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει τέτοια ουσιαστική έκθεση, θα προβεί σε προηγούμενε διαβουλεύσει. Ο εκπρόσωπο τη πολωνική κυβέρνηση μα μίλησε για τη σημασία του άρθρου 22 και τις ανάγκες ε, ενίσχυσης και ανάπτυξή του με βάση τα δικαιώματα που κατοχυρώνει οι συνθήκε. Χρειαζόμαστε επίση και μεγαλύτερη συνοχή, γιατί όλοι συμφωνούμε με την εισηγήτρια ότι ο κόσμο θα πρέπει να ξέρει πού θα αποτανθεί για να λάβει τι πληροφορίε που χρειάζεται. Θέλουμε ένα one-stop shop, να μπορεί από ένα σημείο ενιαία να λαμβάνει πληροφορίε που χρειάζεται, όπου και αν βρίσκεται. Αλλά πρώτα θα πρέπει να συμμαζέψουν τα του οίκου του στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί αυτή τη στιγμή με τον διαμεσολαβητή έχουμε ένα κεντρικό σημείο επαφής. Αλλά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουμε ένα τμήμα για την ελεύθερη διακίνηση και τα, πολιτι... και τα πολιτιακά δικαιώματα, ένα άλλο τμήμα για την κοινωνική ασφάλιση και τα δικαιώματα ασφάλιση, ένα άλλο τμήμα για την αναγνώριση των προσόντων, ένα τέταρτο τμήμα για τα προγράμματα ανταλλαγών που υποτίθεται ότι στηρίζουν αυτή την άσκηση των δικαιωμάτων. Εδώ και καιρό λοιπόν ζητούμε μια μεγαλύτερη συγκέντρωση στο χαρτοφυλάκιο ενό και μόνο επιτρόπου. Γιατί δεν θέλουμε μόνο ο One Shop στην πρόσωψη, θέλουμε και αντίστοιχη κάλυψη, αντίκρισμα από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύτερο συντονισμό. Σε ό,τι αφορά την ε, καλύτερη εφαρμογή, δεν χρειάζεται να μακρηγορήσω γιατί το κάλυψε αυτό εύστοχα η συγγήτρια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, ε, επισημαίνει την ανάγκη λήψης προληπτικών μέτρων για την καλύτερη ε, εφαρμόγη. Όπως είπε και ο κ. Διαμαντουρός, θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση ώστε να καταλάβει ο πολίτης ότι γίνεται σωστή επεξεργασία των ε, αιτιάσεων τους. Ε, θα πρέπει να θεσπιστούν κατάλληλες προθεσμίες, να γίνουν υπόλογα τα θεσμικά όργανα, και φυσικά να διατεθούν και οι αρκετοί πόροι για τη σωστή διαχείριση, επεξεργασία και διεκπαιρέωση όλων αυτών των ε, παραπώνων και των αναφορών. Θα πρέπει επίσης οι πολίτες να αποκτήσουν καλύτερη πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί η πρόσβαση ε, αντιμετωπίζεται ως ε, φυσική απόρρεια της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας. Θα πρέπει λοιπόν να είναι πραγματικά εύκολη η πρόσβαση αυτή των στο δικαστήριο. Σε ό,τι αφορά την περαιτέρω ανάπτυξη ή εμπλουτισμό αυτή τη έννοια τη ευρωπαϊκή ηθαγένεια, πιστεύω ότι θα πρέπει να ξεχνούμε ότι για το θέμα αυτό δεν μπορούμε απλώ να επιβάλλουμε κάποιε διατάξει και να προλάβουμε την κοινή γνώμη, την κρατική θέληση. Παρόλο που Ίσως ε, οι μισοί πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν συνέστηση της ευρωπαϊκής Ιθαγένειας μαζί με την εθνική τους υπηκότητα. Κάτω από τους μισούς ε, θεωρούν ότι είναι μόνο εθνική υπήκοη, έχουν μόνο την εθνική ηθαγένεια. Σε αυτούς τους πολίτες θα πρέπει να φτάσουμε να τους εντάξουμε στη διαδικασία, να βελτιώσουμε την ενημέρωσή τους. Υπάρχει όμως ένα γενικό πλαίσιο για την ανάπτυξη αυτής της έννοιας ευρωπαϊκής Ιθαγένειας και μπορούμε μέχρι χωρίς την συνθήκη της Λισαβόνας να δώσουμε δεσμευτική ισχύ στη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και να πείσουμε την Πολωνική και την Βρετανική κυβέρνηση να αποποιηθούν τις αυτοεξαίρεσεις τους για το Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πρόσβαση στο, στο Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης ως Ένωση. Νομίζω ότι θα πρέπει να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο Τη ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Και εκεί που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δραστηριοθεί περισσότερο και να μην ε, περιορίζεται σε μια πλήση δεξιών αφορών και εκθέσεων είναι να εντοπιστούν κάποιες αδυναμίες σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Για παράδειγμα, όταν οι πολίτε δεν ασκούν ε, επαρκώ το δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγησης στις ευρωεκλογές. Ίσως ε, ε να μην έχουν το δικαίωμα να συμμετέχουν σε εθνικά δημοψηφίσματα στις εθνικές εκλογές και γι' αυτό να μην ασκούν το δικαίωμα συμμετοχής στις εκλογές στη χώρα φιλοξενής, στη χώρα διαμονής. Και με το αντίξω τρέχον οικονομικό κλίμα θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη διάσταση του πολίτη που θα αστερνίζεται και την ευρωπαϊκή αυτή διάσταση. Επίσης θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στην, στα ίσα δικαιώματα όλων των πολιτών, από όποια χώρα και προέρχονται, είναι παλιά χώρα μέλος ή νέα χώρα μέλος. Ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες διευρύσεις του 2004 και το 2007. Στο επόμενο στάδιο θα πρέπει να διαρωτηθούμε μήπως θα πρέπει να αποκαταστήσουμε την ίση μεταχείριση μεταξύ μιας ομάδας μεταναστών που είναι υπήκοοι κρατών μελών και 8,2 εκατομμύρια αυτής της χώρας ζουν σε άλλη χώρα μέλος και διπλάσιος αριθμός αυτών των μεταναστών είναι υπήκοοι τρίτων χωρών, όχι κοινωτικών. Θα πρέπει η ευρωπαϊκή ηθαγένεια είναι μια έννοια που να περιλαμβάνει πολύ περισσότερα, να καλύπτει πολύ περισσότερους πολίτες από ό,τι σήμερα και να κοιτάει και προς τα έξω να μην ενδοσκοπεί Ευχαριστώ θα έλεγα σκέτο τόνι για να μην τα ξανακάνω σαλάτα με το όνομά σας. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν το λόγο. Η Μπάουτενβεχ που είναι υπεύθυνη για την έκθεση εναντίον των διακρίσεων. Κάτε Λάιν έχει το λόγο. Αναρωτιόμουν αν θα έλεγα κάτι για την έκθεσή μου, αλλά τελικά δεν θα πω. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Αναφερθήκατε και στους απάτριδες και η ερώτησή μου αφορά και τους υπόλοιπους εμπειρογνώμονες. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια προέρχεται από την εθνική ηθαγένεια. Πρέπει να έχεις μια εθνική ηθαγένεια από ένα μέλος κράτος και τότε έχεις αυτόματα και την ευρωπαϊκή. Αλλά δεν είναι δυνατόν από ό,τι φαίνεται να είσαι ευρωπαίος πολίτης αν δεν είναι πολίτης κράτους μέλους. Υπάρχουν όμως ορισμένες χώρες και στη Βαλτική, όπου υπάρχουν αρκετοί απάτριδες εκεί. Τι γίνεται. Θα μπορούσε η Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια να διαχωριστεί από την προϋπόθεση σύμφωνα με την οποία για να την έχει κανείς πρέπει να έχει και την ηθαγένεια ενός κράτους μέλους. Πιστεύετε ότι είναι πραγματικά απαραίτητο να έχει κανείς την εθνική ηθαγένεια για να έχει την ευρωπαϊκή. Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Γι' αυτά που είπε ο κύριος Μπιάνκι, προφανώς είναι άδικο για ένα Ιταλό να πηγαίνει στη Δανία, εφόσον δεν έχει βέβαια όλους τους περιορισμούς, αν έχει παντρευτεί κάποιον από το Μαρόκο, τότε κάποιος που ζει στη Δανία και θέλει να παντρευτεί κάποιον από το Μαρόκο δεν μπορεί. Και στην Ολλανδία την ίδια συζήτηση κάνουμε και εμείς έχουμε πιο αυστηρότερη νομοθεσία από κάποιες άλλες χώρες. Φαίνεται ότι είναι λίγο άδικο, αλλά υπάρχει και το θέμα της αμοιβαίας αναγνώρισης. Υπάρχουν διαφορές στα κράτη-μέλη και πρέπει να τις παραδεχθούμε. Ή θα πρέπει να εναρμονίσουμε τα πάντα ή θα πρέπει να δεχθούμε ότι κάποιος ο οποίος πηγαίνει από την Ιταλία στη Δανία και είναι νόμιμα παντρεμένος στην Ιταλία θα θεωρηθεί νόμιμα παντρεμένος και στη Δανία. Δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε επιπλέον προϋποθέσεις και είμαι σαφέστατα υπέρ της αμοιβαίας αναγνώρισης. Νομίζω ότι δεν έχουμε φτάσει βέβαια ακόμα σε αυτό το επίπεδο. Αν δει σαν παράδειγμα το τι γίνεται στην Ολλανδία. Κάποιοι από τους γάμους μας αναγνωρίζονται από άλλες χώρες. Κάποιες άλλες ε, μορφές ένωσης ε, Ολλανδικές, σαν παράδειγμα από ε, το ίδιο φύλλο, δεν γίνονται αντικείμενο αναγνώρισης. Δεν μπορεί οι χώρες να το κάνουν αυτό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι εμείς δεχόμαστε όλους τους λευκούς γάμους αλλά όχι τους μαύρους γάμους. Αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Εμείς δεν έχουμε γάμους για γκέι, ας πούμε για ομοφιλόφιλους στην Ολλανδία. Ένα είδος γάμων έχουμε έτσι κι αλλιώς. Εν πάση περιπτώσει έρχομαι στο τελευταίο σημείο. Υπάρχουν πολλές προτάσεις για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής ηθαγένειας και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει τέτοιες προτάσεις. Όταν βλέπω τι γίνεται στην εσωτερική αγορά διαπιστώνω ότι κάποτε είχαμε ένα πρόγραμμα για την απόσυρση όλων των εμπεδίων και υπήρξε μια όθηση και υπήρξαν τακτικοί έλεγχοι και υπήρξε πρόοδος. Μήπως μπορούμε και στον συγκεκριμένο τομέα σε μία πρώτη φάση να συλλέξουμε τα εμπόδια τα οποία υπάρχουν και να πούμε ότι τα, εμπόδια, τα εμπόδια αυτά θα τα αποσύρουμε, θα τα απομακρύνουμε και για να το πετύχουμε απαιτείται χρόνος. Θα λάβουμε υπόψη μας και κάποια προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν σε τομείς όπως η ασφάλεια κτλ. Και θα πρέπει λοιπόν όπως το είχαμε κάνει και στην εσωτερική αγορά Momentum then. Ε, Ευχαριστώ Κατελάιν για αυτές τις ερωτήσεις προτάσεις. Ποιος θα ήθελε να απαντήσει πρώτος. Ο κύριος Βέναμπλς. Για το τελευταίο σημείο νομίζω ότι οι διαφορές ανάμεσα, που υπήρχαν ανάμεσα στην εσωτερική αγορά είχαν σχέση με το ότι η εσωτερική αγορά ήταν ένα συνεκτικό μέσο διακυβέρνησης οικονομικής ουσιαστικά. Δεν υπάρχει ένας ενιαίος χώρος στα πλαίσια των οποίων, του οποίου μάλλον να εντοπίσει κανείς ε, τα κοινά στοιχεία. Εγώ ήμουνα σε μια επιτροπή με τη Σιμών Βέιε, όπου είχαμε δει ότι χρειαζόντουσαν 85 μέτρα εκείνη την εποχή που έπρεπε να ληφθούν και υπήρχαν πάρα πολλά κενά στην νομοθεσία. Τώρα πια είναι θέμα, όπως λέτε κι εσείς, επιβολής ουσιαστικά. Αλλά απαιτείται ένα ελάχιστο, θα έλεγα, θεσμικής και δικητικής συγκέντρωσης. Και αυτό δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση. Και προσπαθούμε εμείς να ορίσουμε τις ευθύνε έτσι ώστε να εντοπίσουμε σωστά τη σειρά των προβλημάτων που εκκρεμούν. Πάρα πολύ σύντομα για τα τρία αυτά σημεία. Για το αν θα πρέπει να είστε πολίτης μιας χώρας για να είστε πολίτης της Ευρώπης. Εμείς κοιτάμε τη συνθήκη ως έχει σήμερα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Η ευρωπαϊκή ηθαγένεια, η ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη περιλαμβάνει ένα κατάλογο δικαιωμάτων που υπάρχουν στη συνθήκη σήμερα. Δεν θα πρέπει όμως να είναι κανείς πολίτης Ευρωπαίος για να μπορεί να χαίρει των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτά ισχύουν για όλους. Για τη συγκεκριμένη κατάσταση στις συγκεκριμένες χώρες, αυτά θα πρέπει να τα δείτε σε ένα πολύ συγκεκριμένο πλαίσιο, δεν θα πρέπει να γενικεύουμε. Αν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διάφορους λόγους κάποιοι έχαναν την ε, ηθαγένειά τους, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνουν και την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Το ερώτημα αυτό θα μπορούσε να τύχει εξέτασης. Είναι δύσκολο όμως να εφεύρει κανείς νέους κανόνες γιατί η συνθήκη είναι αυτή που είναι. Αυτά που είπα για την αντίστροφη διάκριση δεν εννοώ ότι πρέπει να καταργηθεί. Είναι καλό πράγμα αλλά ταυτόχρονα και επικίνδυνο πράγμα είναι σαν την οικονομική κρίση που δημιουργεί καταστάσεις στα πλαίσια των οποίων είναι δύσκολο για τους πολιτικούς τα κράτη-μέλη να εξηγήσουν τα μέτρα τα οποία παίρνουν. Και αυτό το οποίο συμβαίνει συνήθως είναι να μας ζητούν κάποιοι κανόνες να αλλάξουν, να αποσυρθούν γιατί δεν βολεύουν. Η ιδέα σας, η τρίτη, για να υπάρξει ένας κατάλογος των προτεραιοτήτων είναι κάτι το θετικό για να δούμε πού τα πράγματα πάνε καλά και πού όχι. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Βέναμπολς γιατί κάποια από τα θέματα αυτά είναι τόσο τεχνικά περίπλοκα που να δημιουργήσουμε μία υπηρεσία, μία διεύθυνση είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η κοινωνική ασφάλιση είναι πολύ περίπλοκη, η ελεύθερη διακίνηση είναι πάρα πολύ περίπλοκη επίσης. Πάντως νομίζω ότι σαν ιδέα δεν είναι κακή. Λοιπόν, θα ήθελε κάποιος άλλος το λόγο. Κάσμαν. Καλώς ήρθες. Ε, Συγγνώμη που άργησα και ήρθα την τελευταία ώρα. Είχα άλλη δουλειά, αλλά παρακολούθησα ε, από πολύ κοντά την συζήτηση αυτή για τις αρμοδιότητες και τις συγκρούσεις που παρουσιάζονται κατά την άσκηση δικαιωμάτων ε, της ηθαγένειας και στην Επιτροπή. Υπάρχουν ορισμένες αρμοδιότητες που παραμένουν σε επίπεδο κρατών μελών. Όμως, αν θέλουμε να δώσουμε νόημα στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια, να την κάνουμε μια πραγματικότητα, δεν θα έπρεπε ακόμα και όταν αυτές οι αρμοδιότητες είναι σε επίπεδο κρατών μελών, δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια σειρά δικαιωμάτων που θα ισχύουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αυτό δεν υπάρχει. Η Επιτροπή και οι διερμηνείς έχουν βαρεθεί να με ακούν να εκφράζω αυτή την εμπειρία. Και μάλιστα αυτό δεν έχει να κάνει και με το σεξουαλικό προσανατολισμό. Αλλά αν υπάρχει ας πούμε μια εταιρική σχέση ε, μεταξύ δύο ανθρώπων ή μάλλον ξεχάστε το, ένα ε, δικαίωμα ε, ας πούμε πηγαίνω σε άλλη χώρα που για κάποιο λόγο αυτή η ελεύθερη συμβίωση, η εταιρική σχέση δεν αναγνωρίζεται και είμαι στο νοσοκομείο ανέστητος και χρειάζομαι θεραπεία. Ο σύντροφός μου είναι ο πιο κοντινός μου άνθρωπος, αλλά με βάση την νομοθεσία της άλλης χώρας μέλου δεν θα έχει δικαίωμα. Άρα λοιπόν συρρυκνώνονται τα δικαιώματα κάποιων ανθρώπων ε, και με την εθνότητα έχει σχέση την ε, φίλη, την θρησκεία, τις πεπιθήσεις αλλά και την αναπηρία ως ένα βαθμό. Δεν έχω μιλήσει για το κοινωνικό φύλλο, αλλά φαίνεται ότι και εκεί που υπάρχει αρμοδιότητα κρατών μελών θα έπρεπε να υπάρχει υποχρέωση να τηρούνται κάποια θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα που είναι κοινά σε όλα τα κράτη-μέλη και δεν θα πρέπει να περιορίζονται αυτά από το εθνικό δίκαιο. Ευχαριστώ. Σίγουρα ε, θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Ποιος θα απαντήσει στο Μάικελ που δεν θα αρρωστήσει, επαναλαμβάνω. Συμφωνώ μαζί σας. θα πρέπει να υπάρξουν ελάχιστα επίπεδα προστασίας. Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για τον καθορισμό τους αυτό το οποίο βλέπουμε στην περίπτωση του προγράμματος της Στοκόλμης είναι να προσπαθήσουμε να διανύσουμε τη διάρκεια ζωής τη ζωή ενός ανθρώπου για να βεβαιωθούμε ότι τα δικαιώματά του δεν θα μειωθούν. Ακόμα και σε κάποιον ο οποίος βρίσκεται σε φάση τελική Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει ελευθερία διακίνηση μέχρι τη στιγμή που πεθαίνεις. Από εκείνη τη στιγμή και μετά υπάρχουν ε, εκατοντάδες απαγορεύσεις που δεν επιτρέπουν στο, στη σωρό να ε, επιστρέψει στην χώρα από την οποία προέρχεται. Εν πάση περιπτώσει θα τα δούμε όλα αυτά. Μερικές φορές ε, κάποιοι διεθνείς κανόνες ε, ισχύουν και αρκεί αυτό, άλλες φορές όχι. Πάντως θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι οι προτάσεις τις οποίες θα κάνουμε να είναι ελεγμένες. Σχετικά με ένα χρονοδιάγραμμα εναντίον των διακρίσεων, μεγαλύτερο από αυτό το οποίο προτείνουμε, σε σχετικά με την ελάχιστη σε μέγεθος πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προφανώς κάτι τέτοιο θα είναι χρήσιμο, αλλά απαιτείται και το κατάλληλο φόρουμ. Να πω ότι έχουμε εξετάσει το θέμα των, των γάμων, εν πάση περιπτώσει, ήδη από το 2004 και η ίδια η οδηγία του 2004 η 38 δεν επιβάλλει λύσεις στα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη πολλές φορές δεν σέβονται ούτε τους δικούς τους κανόνες για την αναγνώριση ενώσεων ανθρώπων που προέρχονται από άλλες χώρες. Υπάρχουν πάρα πολλές διαφορές και στρεβλώσεις οι οποίες θα πρέπει να απομακρυνθούν χωρίς να χρειαστεί να φανεί ότι πιέζουμε μια χώρα ή την αναγκάζουμε να αλλάξει την ομοθεσία της. Σε άλλους τομείς του κοινοτικού δικαίου φαίνεται ότι αν μετακινείται κανείς στην Ένωση συνήθως δεν χάνει. Δεν χάνει τη σύνταξή του, δεν χάνει οικονομικά. Γιατί να χάνει σε επίπεδο πολιτικών ελευθεριών όταν μετακινείται από χώρα σε χώρα. Πρέπει να υπάρξει μια ιδέα κεκτημένων δικαίων τα οποία δεν θα πρέπει να αμφισβητούνται. Δεύτερο σημείο. Συμφωνώ με την Επιτροπή ότι δεν θα πρέπει να αποφεύγει κανείς την εξειδίκευση των παραπώνων των πολιτών. Υπάρχουν βέβαια παράπονα στον τομέα της φορολογίας, της κοινωνικής ασφάλισης, του οικογενειακού δικαίου και τελικά μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν θέλετε ένα πρόγραμμα δράσης που να αποσύρει όλα αυτά τα εμπόδια θα πρέπει να υπάρξει μια υψηλού επίπεδου πολιτική ευθύνη που να καθοδηγεί τη διαδικασία να κάνει προτάσεις και στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στα άλλα όργανα. Εγώ δεν λέω λοιπόν ότι όλα θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε μία υπηρεσία αλλά κάπου στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να αναγνωρίζεται μια ξεκάθαρη ευθύνη για το θέμα των ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, ίσως ε, μέσω και της προσπάθειας η χάρτα να γίνει δεσμευτική. Ευχαριστώ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θα ήθελε το λόγο. Um, Δύο πολύ σύντομα σχόλια. Πρώτον, να πω απλώς, γιατί ο διαμεσολαβητής πάντα ήταν υπέρ, ε, υπέρ της αντίληψης των ελάχιστων προτύπων σε πολλούς τομείς, δεν είναι ώρα να τα πούμε αυτά, αλλά πραγματικά αυτός θα ήταν ένας μηχανισμός που πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε, χωρίς να ανταγωνίζεται άλλους τομείς. Ε, δεν, ε, ε, από την άλλη είμαι κατά της ομοιογενοποίησης. με ελάχιστους κανόνες και πρότυπα αποφεύγουμε αυτό το πρόβλημα και αυτό είναι σημαντικό. Δεύτερον, να υπενθυμίσω απλώς ότι σε διαφορετικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά την εσωτερική αγορά η Επιτροπή Κομισιών διατύπωσε πολύ καλή ιδέα που τώρα αρχίζει να δίνει καρπούς Δηλαδή δημιουργήσε τη μικρή μονάδα που λέγεται Solvit και η οποία επιτρέπει άτυπη γρήγορη επίλυση προβλημάτων μέσα σε λίγες εβδομάδες και αν δεν, δίνει αρκετούς καρπούς ε, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η δυναμική του συγκεκριμένου μηχανισμού δεν αναγνωρίζεται παρκώς από τα κράτη-μέλη. Αυτό μπορεί να πάει προς την κατεύθυνση που προτείνει ο κύριος Βέναμπλς και ίσως θα ήταν άξιο να το, θα αξίζει να το εξετάσουμε. Ευχαριστώ όσο έλαβαν μέρος στη δημόσια κρόαση και τους ε, προσκεκλημένους μας από το πάνελ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτριά μας, τη συνάδελφο Ούρσουλα Γκάτσεκ, για τα τελικά συμπεράσματα αυτήν ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων. Ευχαριστώ. Να σας ευχαριστήσω και σας κύριε Πρόεδρε και όλους τους προσκεκλημένους μας. Μερικοί χρειάστηκε να φύγουν γιατί είχαν ανηλυμένες υποχρεώσεις. Άρα νομίζω ήταν πολύ, αυτή και ε, πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση γιατί μιλήσαμε όχι μόνο με την έμπρακτη εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Ιθαγένειας αλλά με κάποια θεμελιώδη της ε, στοιχεία. Για να ανακεφαλαιώσω κάπως τη συζήτηση στην ε, παρουσίαση του κυρίου Σόρα από το Πολωνικό Υπουργείο Εσωτερικών και Διοίκησης της Πολωνίας φάνηκε η ανάγκη μη διακριτικής μεταχείρισης των Ευρωπαίων πολιτών και το θέμα, το, ο προβληματισμός για τους ενδοκινο, ενδοκινοτικούς μετανάστες. Αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή μας, του υπήκου των τρίτων χωρών, οι αιτούντε άσυλο. Πάντως, το τελευταίο χρόνο που είμαι μέρος αυτής της επιτροπή, δεν ασχοληθήκαμε επαρκώσουν αυτά τα θέματα της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης μεταναστών ε, από τη μία χώρα της Ένωσης στην άλλη. Ο καθηγητής Γκαλίτσκι τόνισε στα σχόλιά του ότι δεν είναι μια ιδέα η ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ο Ευρωπαίος πολίτης είναι ένας άνθρωπος με σάρκα και οστά που έχει προβλήματα. Ε, η ανάγκη ενίσχυσης προξενικής προστασίας αναφέρθηκε από πολλούς εμπειρογνώμονες και πάλι στα πλαίσια της κατάργησης διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ των μεταναστών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με βάση και τα δικαιώματα που από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, εκτίμησε ιδιαίτερα τα σχόλια του συναδέλφου από την Κύπρο που ε, δραστηριοποιήθηκε ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα ως συντακτής γνωμοδότησης της ε, Επιτροπής Σταγματικών Υποθέσεων και περιμένω με ανυπομονησία την ε, ισορροπημένη είμαι σίγουρη γνωμοδότησή του γιατί αναφέρθηκε στα κέρια ερωτήματα κατά πόσο γνωρίζουν τα δικαιώματα, τα δικαιώματα τους οι πολίτες και αν όχι γιατί όχι παρόλο που τους, τα δικαιώματα αυτά τους καθιστούν αναπόσπαστο τμήμα της Ένωσης. Είχαμε και τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή μας εδώ, που όταν εμείς κάνουμε κάτι στραβό, εκείνος λαμβάνει τα παράπονα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Μας έδειξε τις ευαισθησίες του και την ανάγκη να σεβαστούμε τις τοπικές ευαισθησίες και να επιδιώξουμε τοπικές θεραπείες και φάρμακα. Επίση, να τονίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Θαγένεια είναι μια προστιθέμενη αξία και συμπληρώνει, δεν υποκαθιστά την Εθνική Θαγέννη. Επίση, ανάγκη μεγαλύτερη διαφάνεια, γιατί πολύ συχνά μιλούμε για τη διαφάνεια στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών. Και ένα από του που οι πολίτες μας αισθάνονται τόσο απομονωμένοι από το έργο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι επειδή δεν καταλαβαίνουν τι συμβαίνει. Θεωρούν ότι όλα γίνονται κρυπτό και παραβίστο και κλεισμένο των θυρών. Όπως σήμερα το πρωί που όλοι περιμέναμε έξω από την αίθουσα για να ολοκληρωθεί η συζήτηση για την τρομοκρατία. Αυτό όμω ήταν εξαίρεση τον κανόνα για λόγου ασφάλεια. Συνήθω οι, ακρα... οι συζητήσει μα είναι ανοιχτέ, είναι δημόσιε και όποιο ενδιαφέρεται μπορεί να τι παρακολουθεί. Άλλωστε η σημερινή δημόσια κρόση αναμεταδιδόταν και από το ίντερνετ, από το web stream. Οπότε είχαμε ε, πολύ μεγαλύτερο ακροατήριο. Έτσι θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών, του οποίου εκπροσωπούμε. Κύριε Μπιάνκι, ήσταν εξαιρετικό για γραφειοκράτη. Γιατί είναι δύσκολο να βρούμε ένα γραφειοκράτη που έχει τέτοια ευαισθησία και επίκριση των προβλημάτων τη εφαρμογή και τη επικοινωνία. Και συγχαρητήρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μα έστειλε τόσο άξιο εκπρόσωπο σήμερα. Είναι σημαντικό να επικεντρωθούμε στο τοπικό επίπεδο. Γιατί οι τοπικές διατάξεις μπορούν να δημιουργήσουν πολλά προβλήματα με αυτούς που μπορεί να διαμένουν σε εργατικές κατοικίες, που μπορούν να εκμεταλλευτούν διάφορα κοινωνικά επιδόματα. Η συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και η συνεργασία με τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή αλλά και τους Εθνικούς Διαμεσολαβητές η ανάγκη αυτής της συνεργασίας φάνηκε και στην δήλωση του Τόνι Βέναμπλς. Το θέμα της προξενικής προστασίας και πάλι. Επισημάνατε κάτι πολύ σημαντικό. Τα κράτη-μέλη δεν είναι και πολύ πρόθυμα για το θέμα αυτό. Και αυτό το καταλαβαίνω για μια χώρα που δαπανά μεγάλο τμήμα του, του ΑΕΠ στις διπλωματικές της υπηρεσίες. Γνωρίζω ότι η Γαλλία έχει ένα τεράστιο προϋπολογισμό για διπλωματικές και προξενικές υπηρεσίες. Οπότε μια τέτοια χώρα μπορεί να πει γιατί να πληρώνουν οι Γάλλοι φορολογούμενοι αυτές τις ε, προξενικές και διπλωματικές αρχές που θα προστατεύουν και υπηκόους άλλων χωρών, που θα εκμεταλλεύονται αυτή την γενναιόδορη παροχή προστασίας. Έχουμε όμως τα περιστατικά της Βομβάης και βλέπουμε να μένουν οι άνθρωποι με τις πιτζάμες τους και να αντιμετωπίζουν μια τρομερή κατάσταση. Και μερικά, μερικοί πρόξενοι δεν έδειξαν ένα στοιχειώδη ανθρωπισμό και μια στοιχειώδη ευαισθησία για τα βάσανα του συνανθρώπου τους. Οπότε το θέμα της χαμηλής συμμετοχής σε ευρωεκλογέ ε, ε, θα είναι την επόμενη φορά περιττό, γιατί θα έχουμε τόσο σημαντική συμμετοχή εξαιτία τη ευαισθητοποίηση των πολιτών, που δεν θα χρειάζεται μια τέτοια έκθεση. Βέβαια, το έργο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να καταργήσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια, αλλά θα πρέπει εμεί οι πολιτικοί να κινήσουμε το ενδιαφέρον των πολιτών. Στην Πολωνία ήδη εγκρίναμε μια νομοθεσία ώστε να είναι διήμερες οι εκλογές, να μπορούν να ψηφίσουν για δύο μέρες οι Πολωνοί, θεωρώντας ότι αυτό θα αυξήσει την ε, συμμετοχή σε εκλογές. Δεν νομίζω πάντως. Μπορεί να βοηθήσει ορισμένες περιπτώσεις, αλλά όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να ψηφίσουν, ακόμη και αν ε, μπορούσαν να το κάνουν με το κινητό τους, δεν θα έμπαιναν στον κόπο, αν δεν ενδιαφέρονταν. Αυτό είναι το δικό μας ε, μέλημα, να κινήσουμε το ενδιαφέρον του πολίτη για να ψηφίσει και εσείς να άρετε τα γραφειοκρατικά εμπόδια. Τα θέματα των διακριτικών μεταχειρήσεων επίσης αναφέρθηκαν εύστοχα. Ο κύριος Βέναβλης με το δύσκολο, πρόφερτο επίθετο είπε ότι το 10 με την ομολογία του χάραξε δρόμο. Θα πρέπει λοιπόν τα κράτη-μέλη να δικαιολογηθούν γιατί ε, θεσπίζουν κάποιους περιορισμούς. Και δεν ε, θα πρέπει οι πολίτες να πρέπει να αποδείξουν ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί. Αναφερθήκατε και στον κύριο Κοχανόφσκι, ο οποίος έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ε, των μεταναστών από τις νέες χώρες μέλη προς τις παλιές. Σίγουρα θα πρέπει να είναι πιο στοχοθετημένη η συζήτησή μας, να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Αυτή ήταν μια μικρή πρόγευση σήμερα η δημόσια μας αυτή ακρόαση της κοινή συζήτηση, αλλά δεν θα πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Το θέμα του One Stop Shop ε, είναι πολύ χρήσιμη πρόταση, αλλά μην ξεχνάτε το γεγονό ότι η πολωνική κυβέρνηση έχει ένα τέτοιο είδο One Stop Shop για τους ε, μετανάστες που επιστρέφουν. Και ήμουν ε, μέλος της Πολωνικής Γερουσίας και χαίρομαι γιατί αυτό το παράδειγμα της Πολωνίας και με τη σχετική σελίδα θα δώσει καλό παράδειγμα και σε άλλες χώρες. Ποιο είναι όμως το κεντρικό θέμα της συζήτησης, ποιο είναι αυτό που μας προβλημάτισε σήμερα. Ο κύριος Κάσμαν πρότεινε να προβλέψουμε κάποιες ε, βασικές προϋποθέσεις, ένα ελάχιστο. Αν όμως ε, ε, καταλήξουμε σε συμβασμό για αυτό το ελάχιστο, θα είναι τόσο ελάχιστο που πραγματικά θα είναι αμεληταίο. Είναι κάτι που είπαν και οι κύριοι Βέναμπλους και Μπιάνκι. Η εθνική ευαισθησία που καθορίζεται από διαφορετικές ταυτότητες μερικές φορές καθιστά δύσκολη την επιβολή ορισμένων διατάξεων στα κράτη-μέλη. Μπορεί να μην μπορούμε να επιβάλλουμε βέβαια κάποιες διατάξεις στα κράτη-μέλη, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να ζητήσουμε να συμμορφωθούμε τις εθνικές τους νομοθεσίες. Αυτό είναι απαραίτητο και μπορούμε να το κάνουμε. Μ' αρέσει αυτή η ιδέα το, της βαθμολογίας κατά κάποιο τρόπο, της σύγκρισης ε, με βάση τους στόχους που θέτουμε. Το θέμα είναι πόσο μακριά μπορούμε να πάμε με την έκθεση μας, πόσο φιλόδοξοι μπορούμε να είμαστε και με την αξιολόγηση της πέμπτης έκθεσης. Πριν γίνει Ευρωβουλευτή ε, κατήρτιζε ε, ένα πρόγραμμα management σε συνεργασία με ιαπωνικές εταιρείες. Ήταν μικρές οι αλλαγέ, αλλά πολύ συχνά αυτό που συμβαίνει σε εταιρείε είναι ότι βλέπουμε ένα τεράστιο πρόβλημα και πανικό να επικρατεί με αποτέλεσμα να μην γίνεται τίποτα. Αυτό που πρότειναν οι Άπωνες και το τελειοποίησαν στις διάφορες γενιές είναι να επιφέρουν κάποιες μικρές αλλαγέ στις εταιρείε τους και να... αυτό το υπόδειγμα θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στη δική μας έκθεση, δηλαδή να θέσουμε σχετικά βραχυπρόθεσμους, απτούς στόχους, προσγειωμένους, γιατί αν θέσουμε μεγαλεπίβουλους, στό, στόχους ε, για τους οποίους δεν θα, μπορούμε να, δεν θα μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε συνένεση, τότε δεν θα κάνουμε τίποτα. Μια τέτοια προσέγγιση λοιπόν με μετριοπαθών ε, και προσγειωμένων στόχων, γιατί στις επιχειρήσεις, στον επιχειρηματικό κύκλο λειτουργεί αυτή η προσέγγιση, γιατί να μην λειτουργήσει και στην πολιτική. Σας ευχαριστώ θερμά για την ε, συμμετοχή. Μερικοί δεν ε, συμμετείχαν στη συζήτηση. Φαντάζομαι η σιωπή τους δηλεί συνένεση με αυτά που υπόθηκαν. Πάντως είμαι σίγουρη ότι θα τροφοδοτήσει τη συζήτηση και θα σας οθήσει να υποβάλλετε και τροπολογία. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ευχάριστη η παρέα των Ευρωβουλευτών και των εμπειρογνωμών και προσκεκλημένων μας. Ευχαριστώ. Τη συνάδελφο Ούρσουλα Γκάτσεκ και ελπίζω να έχει καλή τύχη. Σας ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή σας. Ευχαριστώ την επιμελητία. Τελειώσαμε.